Okay, Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Και παρακαλώ ησυχία στην αίθουσα. Εάν θέλετε να συζητήσετε, παρακαλώ να βγείτε. Έτσι βέβαια πρέπει να είναι πάντα, αλλά σήμερα που έχουμε εδώ την Υπουργό Εμπορίου του Καναδά, πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό τον κανόνα αυστηρά. Σας παρακαλώ λοιπόν, ε, όχι συζητήσεις εντός της αίθουσας. Όπως σας είπα, προσκαλέσαμε την Υπουργό για να συζητήσουμε για την ε, εμπορική συμφωνία με τον Καναδά και ε, δέχθηκε την πρόσκλησή μας. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Οπότε έχουμε σχεδόν μια αίθουσα στην διάθεσή μας για να συζητήσουμε με την Υπουργό για το ΣΥΤΑ, την ε, Συμφωνία για Οικονομικά και Εμπορικά Θέματα. Θα κάνει εισαγωγή η Υπουργό μετά θα δώσω το λόγο στην, στον εισηγητή και τους σκιώδης και μετά και στους υπολείπους. Επειδή ε, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από ό,τι καταλαβαίνω, θα ήθελα παρακαλώ να περιορίσω το χρόνο ομιλία σα στα δύο λεπτά. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε, ο συνήθω, βέβαια, σύντομοι και σαφεί. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Μπέρντ, ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή που διαπίστωσα και από τους συναδέλφους και από εσάς. ευχαριστώ επίσης και τα μέλη της Επιτροπής σας που ήρθαν στην Όταβα πριν από μερικές εβδομάδες. Χαρήκαμε πολύ που ήρθατε στο κοινοβούλιο μα, Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Ε, και θέλω να πω βεβαίω ότι δυστυχώς όσο ήσασταν στον Καναδά έγιναν αυτέ οι απεχθεί επιθέσεις. Εκφράζω την ε, βαθιά συμπαράστασή μου και χαίρομαι που όλοι ε, επιστρέψατε και χαίρομαι που είμαι και πάλι μαζί σας. Ε, είναι για μένα μεγάλη τιμή που απευθύνομαι στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορώ λοιπόν να μιλήσω γαλλικά. Μίλησα γαλλικά και στο Bundestag στο Βερολίνο την προηγούμενη εβδομάδα και εξεπλάγησαν ορισμένοι. Είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ένα από τα πιο σημαντικά κοινοβούλια, μία από τους, ε, ένα από τα πιο σημαντικά δημοκρατικά όργανα στον κόσμο και χαίρομαι πολύ που μπορώ να συζητήσω μαζί σας. Όπως ξέρετε, πολύ πρόσφατα το Βέλγιο συγκλονίστηκε από τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις. Εκφράζω τις βαθύτατες, ε, τα βαθύτατα συλληπιτήριά μου το Καναδά θέλει να εκφράσει την ελληνική του με το Βέλγιο, τους πολίτε του και του κατοίκους των Βρυξελών και είμαστε στο πλευρό σας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Κανένας εταίρος ε, της Ένωσης δεν είναι τόσο συνδεμένος με τις ίδιες αρχές με εσά όπως ο Καναδάς. Κατά τη διάρκεια τη ομιλία μου για την ε, σφαιρική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία θέλω να εκφράσω την ελληνική μαζί σας. Υποθέτω ότι είμαι η πρώτη υπουργό της νέας ε, καναδικής κυβέρνησης που έρχεται εδώ. Έτσι δεν είναι, Μπέρντ. Οπότε να ξεκινήσω με δύο λόγια για την κυβέρνησή μας που εξελέγει τον ε, παρελθόντα Οκτώβριο και ε, το Υπουργικό Συμβούλιο ορκίστηκε στις 4 Νοεμβρίου. Να αναφερθώ σε κάποιες από τις βασικές προτεραιότητές μας και μετά θα μιλήσω λίγο και για τη συμφωνία ΣΥΤΑ και κατόπιν βεβαίως με χαρά να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Η κυβέρνησή μας λοιπόν έχει αναλάβει ως βασική δέσμευση την οποία θα σεβαστούμε διότι ο Πρωθυπουργός μας αυτή τη βδομάδα μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, ε, στα Ηνωμένα Έθνη, για να υπογράψει την ιστορική συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Μία από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησής μας ήταν να διαμορφώσουμε μία ιδιαίτερα πολυάριθμη καναδική αντιπροσωπεία με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων και συγκεκριμένα και των φυλών των ε, ε, αυτοχθόνων που συμμετείχε στην αντιπροσωπεία που πήγε στο Παρίσι. Η δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος είναι βασική θεμελιώδης αξία της κυβέρνησής μας και νομίζω ότι τη συμμεριζόμεθα με την Ευρώπη. Ένα δεύτερο θέμα που είναι και αυτό βασική μας δέσμευση και που θεωρώ ότι πρέπει να αναφέρω σήμερα ενώπιόν σας είναι η αντιμετώπιση του προσφυγικού θέλω να συμμεριστώ με όλους τους Ευρωπαίους ε, την εκτίμηση ότι η κρίση αυτή δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Είναι παγκόσμια κρίση. Και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας δεσμευθήκαμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα αναλάβουμε το μερίδιο ευθύνη. Και δεσμευθήκαμε να δεχθούμε 25.000 ε, πρόσφυγες από τη Συρία στον Καναδά. Ήδη επιτύχαμε στις 29 Φεβρουαρίου αυτόν τον στόχο τονίζω ότι δεν είναι πρόσφυγες που έρχονται στις ακτές μας, στέλνουμε αεροπλάνα στους καταβλισμούς να τους φέρουν στον Καναδά και λαμβάνουν μόνιμη κατοικία προς τον Καναδά και στην πορεία χορήγησης ηθαγένειας και ελπίζω φέτος να φτάσουμε στις 40.000. Αυτό είναι σημαντικό να το μάθετε γιατί ξέρουμε τι σημαντικό θέμα είναι αυτό για την Ευρώπη και θέλω να ξέρετε ότι είμαστε σταθερά στο πλευρό σας όχι μόνο στα λόγια αλλά και στη πράξη. Ένα τρίτο θέμα για το οποίο εγώ είμαι προσωπικά υπερήφανη σε σχέση με την κυβέρνησή μας είμαι πολίτης μιας χώρας ο οποίος ε, είναι υπερήφανος που είναι φεμινιστής. Ο σεβασμός της διαφορετικότητας είναι βασική μας δέσμευση και στις 4 Νοεμβρίου ο Καναδάς απέκτησε την πρώτη κυβέρνηση που έχει 50% άνδρες, 50% γυναίκες υπουργούς. Ναι, γιατί να μην το χειροκροτήσουμε. Είμαι περήφανη για τον Πρωθυπουργό μας που ε, κατήρτισε μια κυβέρνηση με αυτή την ισορροπία φίλων και είναι τιμή, αλλά πραγματικά είναι και πολύ ευχάριστο να συμμετέχει κανείς σε ένα Υπουργικό Συμβούλιο με ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών. Και κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω ως βασική δέσμευση του Καναδά και της νέας μας κυβέρνησης είναι μια βαθιά προσπάθεια για να προωθήσουμε την ε, πολυμερή προσέγγιση. Είμαστε περήφανοι για τον ιστορικό μας ρόλο. Πάντοτε ενθουσιοδός προωθήσαμε τις πολυμερείς μορφές συνεργασίας κάθε είδους. Είναι βαθιά πεποίθηση της κυβέρνησής μας. Ορισμένοι είπαν ότι να, ο Καναδάς επανήλθε στην ε, παγκόσμια σκηνή. Δεν είχαμε αποχωρήσει ποτέ, αλλά ίσως τώρα να συμμετέχουμε λίγο πιο ενεργά στις ε, συναντήσεις για τα παγκόσμια θέματα και στις διεθνείς εταιρικές σχέσεις. Είναι λοιπόν βασική μας αξία, βασική δέσμευση της κυβέρνησής μας. Πραγματικά πιστεύουμε ότι φέρουμε ευθύνη για τον πλανήτη και θεωρούμε ότι η στήριξη των διεθνών θεσμών και μορφών συνεργασίας είναι θεμελιώδης αξία μας και αυτό με φέρνει λοιπόν στην ε, εταιρική μας σχέση με την Ευρώπη που πιστεύω πως θα είναι το βασικό μας θέμα σήμερα. Για μας αυτή η εμπορική συμφωνία με την Ευρώπη είναι για μια σειρά από λόγους ε, ιδιαίτερα σημαντική αλλά ίσως ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι στόχος μας είναι να βαθύνουμε την εταιρική μας σχέση με μια ομάδα χωρών με τις οποίες έχουμε ιδιαίτερα βαθιές κοινέ αξίες. Εδώ αισθανόμαστε στο σπίτι μας και ελπίζω μπέρντε ή και οι συναδελφοί σου να αισθάνθηκαν εξίσου στο σπίτι τους στον Καναδά. Όπως και η Ευρώπη, είμαστε πολυπολιτιστική ε, ενότητα με διάφορες γλώσσες και ε, θέλω να σημειώσω περήφανα ότι ο Καναδάς ανέλαβε την ευθύνη για τη μετάφραση στα γαλλικά τη συμφωνία ΣΥΤΑ και πιστεύουμε στη σημασία Σταθερή οικονομικής ανάπτυξη και καταλαβαίνουμε το ρόλο που παίζουν οι κυβερνήσεις για να προωθήσουν αυτή την οικονομική ανάπτυξη, και για να προστατεύσουν το, τους πολίτες. Έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας ε, που αναλαμβάνει όλα τα έξοδα. Η βασική λοιπόν αξία του ΣΥΤΑ για μας είναι η στενότερη σχέση που αποτελεί με σας σας γουστάρουμε. Πώς να το πω, έχουμε πολλά κοινά. Και θεωρούμε ότι έχει μεγάλη αξία η πιο στενή συνεργασία μαζί σας. Και στη σχέση μαζί σας, αλλά και ευρύτερα για τον κόσμο. Κάτι άλλο που επίσης θέλω να τονίσω σε σχέση με τη Συμφωνία ΣΥΤΑ είναι η σημασία που μπορεί να έχει αυτή η συμφωνία για να προκύψει οικονομική ανάπτυξη. Αναφέρθηκα στις αξίες της κυβέρνησής μας. Αλλά όπως και εσείς, είμαι εκλεγμένος εκπρόσωπος. Κατά την προεκλογική στρατεία, το βασικό θέμα που τέθηκε είναι η στασιμότητα στην οικονομία και οι φόβοι των μεσαίων τάξεων για το εισόδημα και την απασχόλησή τους. Αυτή είναι η βασική μέρημνά μας ως κυβέρνηση και εγώ ως προοδευτική πολιτικός ανησυχώ γι' αυτό. Εάν δεν επανέλθει η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους υπόλοιπους στόχους μας. Για το περιβάλλον, στον Καναδά ένα βασικό θέμα είναι οι κοινότητες αυτοχθόνων που έχουμε και θέλουμε να υπάρξουν οι αναγκαίε δαπάνε για να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και περίθαλψή του. Όλοι αυτοί οι στόχοι χρειάζονται οικονομική ανάπτυξη και η ΣΥΤΑ θα παίξει μεγάλο ρόλο ως κίνητρο για την οικονομική μας ανάπτυξη. Σε μια κοινή μελέτη που εκπονήσαμε μαζί από το 2008 και επειδή ορισμένες συμφωνίες του ΠΟΕ δεν επετεύχθησαν που τότε θεωρούσαμε ότι θα έχουν επιτευχθεί. Αλλά σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη συντηρητική λοιπόν εκτίμηση λόγω του ότι όλες οι προϋποθέσεις δεν έχουν ε, εκπληρωθεί αυτή η συμφωνία θα αυξήσει κατά 23% τις εμπορικέ μας συναλλαγές. Όταν εφαρμοστεί πλήρω, θα αυξήσει το ΑΕΠ μας κατά 0,77% ετησίω. Αυτή είναι σημαντική ε, όθηση για την οικονομία. Αυτό σημαίνει Περισσότερε δουλειέ, περισσότερο εισόδημα για τους εργαζόμενους. Και κάτι ακόμη. Και τελευταίο. Γιατί νομίζω ότι όλοι το έχετε πολύ κατά νου και ενδεχόμενα το έχετε συζητήσει. Υπήρξε μία πολύ σε βάθος νομική εξέταση του κειμένου. Νομική επαλήθευση. Η... Το κόμμα μας υποστήριξε αυτή τη συμφωνία και όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση. Αλλά όταν ε, κάναμε κυβέρνηση, ξέραμε κάποιες ανησυχίες των Ευρωπαίων για το κεφάλαιο για τις επενδύσεις. Και νομίζω ότι εξεπλάγησαν λίγο οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, διότι η νέα κυβέρνηση, αντί να θεωρήσει ότι οι ευρωπαϊκές απαιτήσει για το θέμα αυτό ήταν πρόβλημα, συμφωνήσαμε. η κυβέρνησή μου και εγώ προσωπικά είμαστε προοδευτική κυβέρνηση. Οπότε είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την εργασία που επιτελέσαμε μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για να διευκρινιστεί το θέμα του κεφαλαίου για τις επενδύσεις. Με μια νέα προσέγγιση. Είναι μια νέα προσέγγιση για ένα κεφάλαιο επενδύσεων σε εμπορική συμφωνία. Διότι προβλέπει τις κατάλληλες αυξημένες αρμοδιότητες που έχει ένα δημοκρατικά εκλεγμένο, μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση για να ελέγχει τις επενδύσεις. Τονίζουμε λοιπόν το ρόλο της κυβέρνησης και νομίζουμε ότι αυτό είναι σωστό και χαίρομαι που το επιτύχαμε μαζί. Επίσης, είναι πολύ μεγαλύτερη η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα και ο ηθικός χαρακτήρας, θα έλεγα, της διαδικασίας επίλυσης διαφορών. Και όσοι ανησυχούν, και ξέρω ότι κάποιοι σε αυτό το χώρο μπορεί να ανησυχούν και εγώ μπορεί να συμμερίζομαι σε ένα βαθμό τι ανησυχίε του για τι εμπορικέ συμφωνίε γενικά. Για το εάν και κατά πόσο οι εμπορικέ συμφωνίε είναι πάντα προ το συμφέρον των λαών. Θα ήθελα λοιπόν να πω για αυτέ τι ανησυχίε η συμφωνία αυτή μεταξύ του Καναδά και της Ένωσης θα είναι πραγματικά πρότυπο. Θα θέση υψηλότερα τον πύχη για προοδευτικές εμπορικές συμφωνίες διεθνώς. Και φυσικά έπρεπε και οι δύο να συμβάλλουμε, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει κάποιες απόψεις για να βελτιώσει μια εμπορική συμφωνία, αλλά πρέπει να υπάρξει συμφωνία για να εφαρμοστούν αυτές οι νέες ιδέες, να δημιουργηθούν νέα προηγούμενα, να δημιουργηθεί ένα νέο επίπεδο φιλοδοξίας. Αυτό ισχύει σίγουρα για μας τον Καναδά, μερικές από τις νέες προοδευτικές διατάξεις στη ΣΥΤΑ είναι για μας μεγάλης αξίας και θα συνεχίσουμε από κοινού με την Ευρώπη διεθνώς να τις προωθούμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, συμπεριληφθούν στις ε, άλλες εμπορικές συμφωνίες που έχουμε όσο θα τις αναθεωρούμε και εξυγχρονίζουμε. Είμαι λοιπόν υπερήφανη για αυτή τη συμφωνία. Νομίζω ότι θα δημιουργήσει περισσότερη ευημερία για όλου, περισσότερε ευκαιρίε για οικονομική συνεργασία μεταξύ του Καναδά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε τομεί κλειδί, ιδιαίτερα για το περιβάλλον, για καθαρέ τεχνολογίε. Στο Βερολίνο έκανα μια συνάντηση στο Δημαρχείο την προηγούμενη εβδομάδα και είδα πόσε καναδικέ συμφωνίε εργάζονται για καθαρέ τεχνολογίε και πραγματικά είναι υπέρ του ΣΥΤΑ γιατί υπάρχει πολύ ευρωπαϊκή τεχνογνωσία στον τομέα αυτό αλλά πάνω απ' όλα είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που μπορώ να τα συζητήσω αυτά μαζί σας γιατί αυτή η συμφωνία είναι μια βαθιά στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της χώρας μου και της Ένωσης που βασίζεται σε αξίες που συμμεριζόμεθα ολόψυχα. Ευχαριστώ και να απαντήσω τώρα σε ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Να δώσουμε τώρα τον λόγο στον εισηγητή και τους πιο δυσηγητές για τον Καναδά και μετά στα υπόλοιπα μέλη. Έχουμε 25 λεπτά για ερωτήσεις και μετά φυσικά θα απαντήσει και ο Υπουργός. Όλα στο τέλος. Ναι, ναι, νομίζω ε, δεν θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε το χρόνο. Παρακαλώ λοιπόν ε, ε, να τηρήσετε το όριο των δύο λεπτών, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε πολλά από τα μέλη της Επιτροπής. Ο εισηγητής, ο κύριος Παπρίξ δεν είναι εδώ. Ο κύριος ε, Κασπαρή από το ΕΛΚ θα τον αντικαταστήσει. Δύο λεπτά. Κατά τη γνώμη μας, το ΣΥΤΑ είναι θαυμάσια συμφωνία Έλεγα λοιπόν είναι πολύ καλή συμφωνία. Αν δει κανεί τι γίνεται για τους δείκτες προέλευσης, για τα τελωνία, ο τομέας της προστασίας των επενδύσεων έχει βελτιωθεί και σας ευχαριστούμε όλοι και νομίζω ότι πρέπει να τεθεί το ερώτημα για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο πρώτος μας εταίρος αν δεν είναι ο Καναδάς. Είμαστε και οι δύο λειτουργούν τα δημοκρατικά συστήματα, ε, ε, είμαστε στην πρωτοπορία της προστασίας του περιβάλλοντος και γι' αυτό θέλουμε να προχωρήσει. Και το δεύτερον, εδώ και 1,5 χρόνο είναι στο ίντερνετ το κείμενο. Και δεν είδα καμία επίκριση για το κείμενο αυτό μέχρι τώρα. Θα έπρεπε και θέλω το επόμενο εξάμεινο η κοινή γνώμη να μπορέσει να εξετάσει το κείμενο αυτό. Θα υπάρξουν και μεταφράσεις Νομίζω ότι είναι όριμη τώρα η συμφωνία. Πρέπει να ξεκινήσει βεβαίω με το σωστό τρόπο, αλλά όσο δυνατόν ταχύτερα η διαδικασία επικύρωση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό να προχωρήσουμε. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμη με την παρουσία σα και θα ήθελα να παραμείνουμε σε επαφή κατά τη διάρκεια τη διαδικασία. Ε, ε, να είμαστε σε επαφή κατά τη διάρκεια τη διαδικασία επικύρωση. Ο εισηγητή και των σελστών δεν είναι εδώ. Ο κύριο David Μάρτιν θα τον αντικαταστήσει. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον Ντάνελ. Πρόκειται για φιλόδοξη και σημαντική συμφωνία και για τις δύο πλευρές. Ε, χαίρομαι που καταφέραμε να έχουμε και μία ε, συμφωνία για τις δημόσιες ε, συμβάσεις και επίσης ε, έχουμε και συμφωνία στα 4GI, στο Αργιουλής, δεν ξέρω αν ακούει η Αμερική, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και θέλουμε να τα συμπεριλάβουμε και στην TTIP. Ε, χαίρομαι ε, για τα όσα είπατε για την αλλαγή του κεφαλαίου για τις επενδύσεις και ότι ο Καναδάς ε, είναι διατεθειμένος να περάσει σε ένα ε, καινούριο σύστημα επενδύσεων. Η πολιτική μου ομάδα δεν τα έχει ε, μελετήσει. είμαστε πολύ ευχαριστημένοι όμως. Αν δεν είχε αλήξει το σύστημα ISDS της επίλυσης των διαφορών δεν θα είχαμε υπερψηφίσει τη συμφωνία και θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, τι γίνεται με την εμπειρία σας ε, στον Καναδά, με την ναύτα και ε, από την εμπειρία αυτή θεωρείτε ότι είναι καλό το νέο σύστημα. Πιστεύετε ότι θα σταματήσει τις ανέτειες αγωγές και μήπως οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τον Καναδά ως παραθυράκι για να κάνουν αγωγές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάτι ακόμα, το συζητήσαμε εμεί το γεύμα, αλλά θα ήθελα να το πω και για την Επιτροπή. Για τα δύο πράγματα που δεν συζητήσατε, για τι συλλογικέ συμβάσει και την παιδική εργασία, μπορείτε να μα εξασφαλίσετε ότι περάτε, περνάτε προ την κύρωση από πλευρά Καναδά. Και τέλο, κάτι πιο προσωπικό. Ξέρετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν νομίζω ότι θα συμβεί, αλλά εάν φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο Πιστεύετε ότι υποτιμούμε την, ε, και θα υποσκάψει αυτό τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ΣΥΤΑ με τον Καναδά. Η κυρία Μακλάρκινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ που είστε εδώ σήμερα. Χαιρόμαστε που έρχεστε εδώ να μιλήσετε με τους βουλευτές και να συνεχίσετε το διάλογο που έχουμε ξεκινήσει για τη ΣΥΤΑ. Και θα ήθελα να σας επενέσω και για τα όσα κάνατε και εσείς και η Σεσίλια Βάλστρομ, δύο ισχυρές γυναίκες ε, ε, και τα όσα έχετε κάνει για να φροντίσετε να προχωρήσει η ΣΥΤΑ και να έχουμε αποτελέσματα. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να έχουμε εμπορικές συμφωνίες που ανοίγουν περισσότερες ευκαιρίες για τις χώρες μας. Και ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ώστε πραγματικά να απολαμβάνουμε και οι δύο τα ωφέλη. Ε, κάποιοι μπορεί να μην εκτιμούν ε, το γεγονός ότι ξανανοίξατε μια ε, διαπραγμάτευση που είχε ολοκληρωθεί. Σταματάει και το κατεστημένο εδώ. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχει κλείσει, είναι πλέον οι 10 εντολές, έχετε ξεκινήσει την εφαρμογή με την κυβέρνησή σας ώστε η κύρωση να προχωρήσει. Ευχαριστώ για τους φιλελευθέρους. Τώρα η κυρία Σάκε. Σας ευχαριστώ. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την πρόσφατη επίσκεψή μας στον Καναδά και να επαναλάβω κι εγώ ότι πραγματικά ήταν πολύ θερμή υποδοχή ε, στον Καναδά τον περασμένο μήνα. Νιώσαμε σας στο σπίτι μας και νομίζω ότι έχει ε, εμβαθύνει και τη δέσμευσή μας για μεγαλύτερη και καλύτερη εμπορική ε, εταιρική σχέση. Ε, νομίζω ότι αυτά τα οποία έχουν προχωρήσει στη ΣΥΤ είναι καλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε από του διάφορου ενδιαφερομένου στον Καναδά τι θεωρούν αυτοί ότι είναι σημαντικό, κυρίω τη διαφοροποίηση του εμπορίου και να μην εξαρτώνται τόσο πολύ από τι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά να μπορέσουν να ενισχύσουν και του δεσμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό που το ακούσαμε από του ίδιου του επιχειρηματίε και επίσης ε, και την ζωτικότητα και τη σημασία της συμμαχίας μας. Μας συγκίνησε, πρέπει να πω, η ε, υποδοχή από όλους, από τους πανεπιστημιακούς, τους φοιτητές, ε, στο στάδιο του χόκι, ε, επιχειρηματίες, άνθρωποι που πραγματικά ένιωσαν βαθιά λύπη μετά από τις επιθέσεις της Βρυξέλλες και μας μεταβίβασαν αυτό το μήνυμα, τήρησαν ενός λεπτού σιγή και απότισαν και φόρο τιμής με διάφορους τρόπους θα ήθελα να συγχαρώ και εσά και τον Πρωθυπουργό Τριοντό και το υπόλοιπο Υπουργικό σα Συμβούλιο για την πραγματικά προοδευτική σα ηγεσία. Είναι τόσο ανανεωτικό, ακούγοντα και τον τόνο των ε, προεκλογικών δηλώσεων στι Ηνωμένε Πολιτείε και την όλη συζήτηση όχι μόνο για το εμπόριο, αλλά στην Ευρώπη και για άλλα θέματα, όπω και το προσφυγικό. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια πολύ καλή στιγμή και πρέπει και εμεί να την επωφεληθούμε από αυτή την ορμή. Και εσεί ω ε, κυβέρνηση Έχετε άρει ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο, το θέμα της, ε, των προστατευόμενων και το κεφάλαιο αυτό και είναι πολύ καλό αυτό και θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε και για μας. Ε, η πολιτική μας ομάδα ελπίζει ότι οι πολίτες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μεγαλύτερες ε, επιχειρήσεις θα αρχίσουν σύντομα να βλέπουν τα ωφέλη αυτής της τόσο σημαντικής συμφωνίας και εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα φροντίσουμε η συμφωνία να έχει αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν. Θα ήθελα να ακούσω και την εντύπωσή σας σε σχέση με άλλους ε, ευρωπαϊκούς φορείς με τους οποίους ήρθατε σε επαφή, κυρίως από κράτη-μέλη. Άκουσα απειλή, βέτο από τους Ρουμάνους φίλους μας και θα ήθελα να ξέρω ε, αν νομίζω ότι υπάρχει κάποια σε αυτό. Ευχαριστώ για την ε, Γκουή κυρία Μινά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Κύριε Υπουργέ, κύριε Φρίλαντ, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Χαιρόμαστε που η φωνή μας ακούγεται στον Καναδά. Εγώ προέρχομαι από την Ενωτική Αριστερά. Ε, είναι η μόνη ομάδα που έχει ίσο, ανδρο, ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών στη σύνθεσή της το έργο που σας περιμένει στην διαπραγμάτευση συμφωνία ΣΥΤΑ είναι δύσκολο, θα είναι δύσκολο, δυσχερές για σας. Ε, θέλουμε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια. Ακούγονται πολλές κριτικές για τη συμφωνία. Η συμφωνία αυτή δεν είναι καλή για τους πολίτες ούτε του Καναδά ούτε της Ευρώπης. Είναι καλή για τις πολυεθνικές. Ε, αυτές ικανοποιήθηκαν, αυτών οι επιθυμίες ικανοποιήθηκαν. Το ίδιο και με την ISDS. Με το, μέσο του ISDS εννοώ, του συστήματος ε, πύλης διαφορών, ε, Ε, γνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι αυτό το σύστημα από την αυτά. Ε, θα είναι και πάρα πολύ κοστοβόρο άλλωστε. Το σύστημα ISDS αφαιρεί αρμοδιότητες και την δυνατότητα να νομοθετούμε και εμείς και ο Καναδάς. Ε, αναφέρεται ότι θα μπει σε εφαρμή το 2017 πολύ πριν τα κράτη-μέλη ε, ε, ακούσουν τη γνώμη των πολιτών τους. Γιατί δεν περιμένετε να λειτουργήσει η δημοκρατική διαδικασία πρώτα. Ευχαριστώ και ο Ζαντό. Και εγώ είμαι πολύ φεμινιστής, οπότε... Αλλά ε, ε έχω και κάποια όρια που μου επιβάλλει το σώμα μου που ακόμα δεν έχω ξεπεράσει. Κύριε Υπουργέ, πράγματι στο ε, παγκόσμιο πολιτικό στερέωμα είναι, μια, είναι φρέσκος αέρας αυτός που φέρατε εσείς με την κυβέρνησή σας και η σύνθεση της κυβέρνησης και αυτό που μας φέρνει. Ε, και ο, ο φιλελευθερισμός της και η προοδευτικότητά της. Ε, βέβαια, για μένα αυτό περιορίζει την, ε, ε, το περιεχόμενο, δηλαδή ε, να πούμε ότι οι συμφωνίες ελεύθερων, ελεύθερων εμπορίου ε, πάντοτε και χωρίς όρους ε, βελτιώνουν την απασχόληση, την ανάπτυξη κλπ. Δεν είναι σωστό. Υπάρχουν κάποιοι τομείς που ευνοούνται, που ωφελούνται, κάποιοι που υποφέρουν, το ίδιο και με τα τμήματα του πληθυσμού. Ε, πιστεύω ότι θα έπρεπε να το αντιληφθούμε αυτό. τώρα, Πιο συγκεκριμένα, μιλήσατε για την επενδυτική συμφωνία. Ε, ακούω ότι το ISCS είναι καλύτερο από το ISDS σε περιφορών. Όμως εγώ δεν έχω δει ούτε ένα επιχείρημα που να ε, επιβεβαιώνει ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο σύστημα επίλυσης διαφορών πέραν των εθνικών ε, δικαστικών συστημάτων. Ε, δεν άκουσα κανένα παράπονο από καναδική εταιρεία για, για την κατάσταση δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε και το αντίστροφο. Ε, η Τρανς ζητά 15 εκατομμύρια δολάρια αποσημείωση από τις ΗΠΑ γιατί ο Ομπάμα αποφάσισε να πολεμήσει την κλιματική αλλαγή ε, παίρνοντας συγκεκριμένα μέτρα τα οποία την έθιξαν ε, για την υγεία για παράδειγμα η συμφωνία αυτή θα επηρεάσει ε, το, την ημί των φαρμάκων ε, και μάλιστα εσείς είδατε, εσείς αποφάσισατε να πάρετε μέτρα για να αντιμετωπίσετε αυτή την αύξηση των φαρμάκων με επιδοτήσεις ε, ε, πρόεδρος. Now we have... Μετά τους και ηγητές περνάμε στους υπόλοιπους ομιλητές, Επτά στον αριθμό, Δύο λεπτά στον καθένα παρακαλώ. κυρία Μασκά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ ε, χαίρομαι που δόθηκε σε μια γυναίκα η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εμπορίου. Ελπίζουμε ότι αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να λάβουμε υπόψη τη διάσταση του φύλου και σε ένα θέμα το οποίο μέχρι τώρα ε, δεν έχει απασχολήσει καμία γυναίκα, όπως έκανε και ο ΠΟΕ τον περασμένο Οκτώβριο. Η μία ερώτηση πέραν της ε, συμφωνίας ε, της ΣΕΤΑ αφορά το καθεστώς οικονομίας της αγοράς προς την Κίνα. Κατά την άποψή μα, από ό,τι γνωρίζουμε, η καναδική κυβέρνηση είπε ότι είναι αντίθετη στο καθεστώ αυτό και χρησιμοποιεί διαφορετική ε, μεθοδολογία για να υπολογίσει την καταπολέμηση του ντάμπινγκ. Η ερώτηση μου είναι εξή. Θα θέλαμε να ξέρουμε τι νομικέ ε, συνέπειε ε, θα υπάρχουν σε σχέση με αυτή την εναλλακτική μεθοδολογία υπολογισμού των μέτρων καταπολέμηση του ντάμπινγκ και κατά πόσον η καναδική κυβέρνηση έχει κάνει και διαβουλευσει με του μεγαλύτερου τους εταίρους, τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Ευρώπη, για το πώς θα πρέπει να διαχειριστεί το ζήτημα στα πλαίσια του ΠΟΕ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρένα, παρακαλώ. Ε, το γεγονός ότι επικρίνουμε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεν σημαίνει ότι δεν μας αρέσει ο Καναδάς. Ε, το ίδιο και με τις ΗΠΑ. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ του αυτά δύο πράγματα. Ε, γιατί Μερικές φορές όταν επικρίνουμε κάτι δημιουργούμε την εντύπωση ότι ε, δεν μας αρέσουν οι κάτοικοι της συγκεκριμένης χώρας ή ε, διαφωνούμε μαζί τους. Ε, μετά τα όσα είπε και ο Ζαντό, σε ό,τι αφορά το ICS, αυτή τη στιγμή επικρίνεται το ICS ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα από τους Γερμανούς δικαστές που λένε ότι αυτό το σύστημα δεν είναι διεθνές δικαστήριο ε, εσείς πώς το βλέπετε το θέμα αυτό. Δεύτερον για το ICS πάλι. Εσείς ε, έχετε κάποιες, ε, κάποια παράπονα για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη που να σας οδηγούν στο να ζητάτε το, την εφαρμογή του ICS. Υπάρχει μια τέτοια δικαιολογία, υπάρχει κάποιος τέτοιος λόγος για την ύπαρξη του ICS. Δεύτερον, για τις, αυτό που σας συνδέει με την Ευρώπη. Ασφαλώς έχουμε πολύ κοινά στάνταρ, αλλά είσαστε πολύ πιο πολύ πιο κοινά στάνταρ με τις ΗΠΑ. Πάνω από 40.000 αμερικανικές επιχειρήσεις είναι εγκαταστημένε στον Καναδά. Ε, μήπως ε, η ΣΥΤΑ θα ανοίξει το παράθυρο στις αμερικανικές αυτές επιχειρήσει ε, για την Ευρώπη. Τρίτον, λέτε ότι θα αποτελέσει παράδειγμα αυτή η συμφωνία. Εγώ έχω κάποια προβλήματα. Για παράδειγμα, με τις θετικέ και τις αρνητικές, ε, τους αρνητικούς και θετικού καταλόγους. Στον ΠΟΕ, ε, ως τώρα έχουμε λειτουργήσει με θετικού καταλόγους, δηλαδή απελευθέρωνουμε, ρώνουμε εκτό και αν. εσεί με συντηρητική κυβέρνηση αποφασίσατε να δουλέψετε με αρνητικού καταλόγους, δηλαδή... Ε, με εξαιρέσει από την απελευθέρωση. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο ε, υποστηρίζετε αυτό το μοντέλο απελευθέρωση. Thanks very much. Um, and thank... Darling, ευχαριστώ για την ομιλία σας. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ στις Βρυξέλλες. Τα είχαμε πει και στην Ότοβα. Η Μαρίτια επίσης ε, μίλησε εκ μέρους αντιπροσωπείας. Σας ευχαριστούμε για την στήριξη που μας έδωσαν όλοι οι Καναδοί συνάδελφοι και εσείς μετά τις επιθέσεις της Βρυξέλλες. Ήταν ε, ιδιαίτερα δύσκολο να είναι κανείς μακριά από το σπίτι του σε τέτοια συγκυρία. Όλοι όσοι ήταν στην ε, αντιπροσωπεία και πιο συγκεκριμένα αυτοί που ήταν συναντήσει, που ήταν περισσότεροι από τα μέλη τη αντιπροσωπεία, γνωρίζουν την ενεργητικότητά σα, τον ενθουσιασμό σα, την αποτελεσματικότητά σα για να προκύψει η ΣΥΤΕ, να επικυρωθεί. Αλλά άλλοι στην Ένωση, αλλά και στο Καναδά, τα βλέπουν λίγο διαφορετικά. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη εκφράστηκαν ανησυχίε για τις δημόσιες υπηρεσίες, για την αναθεωρημένη διαδικασία επίλυσης διαφορών, για τα δικαιώματα των εργαζομένων και αυτές τι ανησυχίε τις διαπιστώνουμε και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού γιατί συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους τη κοινωνία των πολιτών και των συνδικάτων και εκεί και εδώ. Επιπλέον, ορισμένα στοιχεία αυτής της συμφωνίας ανησυχούν περισσότερο τους Καναδούς θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε την άποψή σας επ' αυτού. Γιατί είναι κάπως ε, μονομερής η συμφωνία. Για παράδειγμα, η παράταση του χρόνου προστασίας για τα φάρμακα ε, προστασίας ε, της ε, σύστασης. Yes. Το διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τα φάρμακα. Αυτό θα βοηθούσε τις ε, ε, μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Έχετε εθνικό σύστημα υγείας, αλλά δεν έχετε εθνικό σύστημα παραγωγής φαρμάκων. Δεν σας ανησυχεί αυτό, επειδή υπάρχει και γύρανση του πληθυσμού. <laughs> Ναι, ε, Ο κύριος ε, Φέλια. Φιέλνα. Σας ε, καλωσορίζουμε εδώ. Μα είναι τόσο καταπληκτικό που συμφώνησαν ε, οι δύο αυτοί εταίροι για μια συμφωνία. Αν εμεί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον Καναδά, με ποιον θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Χαίρομαι που θα είναι σε βάθος και σφαιρική αυτή η συμφωνία, νέο πρότυπο για εμπορικές συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες παντού. Αλλά κάτι που με ανησυχεί όχι στην ίδια τη συμφωνία, αλλά στον τρόπο με τον οποίο ε, συνήφθη. Γιατί τι είναι το πρόβλημα. Συμφωνήσαμε σε κάτι, ε, κάναμε και το νομικό έλεγχο και μετά είπαμε «Α, πρέπει να θεωρήσουμε ορισμένες διατάξεις». Γιατί εγώ άκουσα τόσους ε, Καναδούς εκπροσώπους που λένε όχι όχι δεν είναι λανθασμένα αυτά μην τα αλλάξετε. Αφού έχουμε καλό σύστημα για την επίλυση διαφορών ISDS γιατί να το αλλάξουμε για κάτι που δεν ξέρουμε πώ λειτουργεί. Και ξαφνικά αλλάξατε άποψη. Και αυτό νομίζω ότι κάνει κακό στη φήμη του Καναδά. Αλλά το, το γεγονό ότι ξανανοίξαμε θέματα μετά το νομικό έλεγχο είναι κακό και για μας. Αντίθετα με ορισμένου, Εγώ ελπίζω οι αμερικανικέ εταιρείε να μπορέσουν να ωφεληθούν από αυτή τη συμφωνία για να μα προσφέρουν υπηρεσίε. Αν οι αμερικανικέ εταιρείε, οι εταιρείε των ΗΠΑ, είναι διατεθειμένε να σεβαστούν τα υψηλότατα πρότυπα που προβλέπει αυτή η συμφωνία, γιατί όχι. Γιατί η εντύπωσή μου είναι ότι η ΣΥΤΑ είναι πολύ ευρύτερη, πάει πολύ παραπέρα από την ναύτα. Μπορείτε παρακαλώ να μας εξηγήσετε μερικές από τις διαφορές ΣΥΤΑ και ναύτα. Σούστα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Χαίρομαι για την παρουσία σας. Χαίρομαι που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Αυτό αποδεικνύει ότι όντως είναι ιδιαίτερες και πολύ καλές σχέσεις Ένωσης Ευρώπης. Συγγνώμη, Ένωσης Καναδά. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ε, σοβαρά προβλήματα. Γιατί τώρα που κλείνει η συμφωνία, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση που αφορά σημαντικά τμήματα της συμφωνίας. Βεβαίως, μετά τις αλλαγές της συμφωνίας υπάρχουν μερικά πολύ επίμαχα θέματα για μας εδώ στην Ευρώπη. Θέματα που δεν είναι εύκολο να περάσουν. Για παράδειγμα, το νέο σύστημα προστασίας των επενδύσεων. Θέτει πολλά θέματα. Είναι όντως έτσι όπως, όπως το θέλαμε. Υπάρχει μια ευρεία συζήτηση. Χρειαζόμαστε τέτοιε ειδικέ δικαιοδοσίε όταν οι εταίροι έχουν πολύ υψηλά, υψηλά ανεπτυγμένο, ιδιαίτερα ανεπτυγμένο δικαστικό σύστημα. Γιατί χρειαζόμαστε αυτές τις ε, διατάξεις stand still. Διότι έχουμε τις συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εργασίας που καλύπτουν αυτά τα θέματα. Τίθενται λοιπόν μερικά βασικά θέματα. Ξέρω ότι ε, δεν έχουμε συνήθως τόσο πολλές επιφυλάξεις, αλλά λόγω των ιδιαίτερων σχέσεων πρέπει να τα θέσουμε. Θα είχε λοιπόν έννοια ε, να υπάρξει περαιτέρω συμπλήρωση του κειμένου κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις. Γιατί νομίζω ότι ορισμένα τμήματα έτσι όπως είναι διατυπωμένα τώρα θα δημιουργήσουν πολλές αντιδράσεις. Ανέφερα συγκεκριμένους τομείς. Υπάρχει διάθεση να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Γιατί οι επικρίσεις άρχισαν στην Ευρώπη όταν ε, τα βασικά σημεία της συμφωνίας είχαν ήδη συμφωνηθεί. Ήταν κακή η ε, αλληλουχία. Ευχαριστώ η Καρολίν. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Χαίρομαι που κάνατε τόσο δρόμο για να έρθετε εδώ. Σημερίζομαι κάποιες επιφυλάξεις. Σε ορισμένους τομείς ε, διαπιστώνουμε προβλήματα, ανησυχίες των πολιτών που πρέπει να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη. Έγινε κάποια βελτίωση στο κεφάλαιο ISDS, ήταν ένα πρώτο βήμα, αλλά το Φεβρουάριο ακούσαμε ότι δεν θα θυγούν άλλα κεφάλαια. Οπότε η ερώτησή μου, σε τελευταία ανάλυση, θα πρέπει να αποφασίσει ναι ή όχι το Κοινοβούλιο. Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει τρίτη δυνατότητα, δηλαδή κάποια κεφάλαια που δημιουργούν ανησυχίες, αφιβολίες, να τα ανοίξουμε και να τα βελτιώσουμε. Υπάρχει λοιπόν τρίτος δρόμος. Να μην είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ναι ή όχι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας ευχαριστω πολυ ευχαριστω ευχαριστω κυριε ε, Υπουργέ και σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Δεν ήμουν εγώ στην αντιπροσωπεία στον Καναδά, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πραγματικά μεταδίδεται ενέργεια, θάρρος και αποφασιστικότητα. Ως υπεύθυνη για θέματα φύλου ε, από πλευράς των σοσιαλιστών εδώ στην Επιτροπή μας, χαίρομαι που ο Καναδάς έχει μια κυβέρνηση όπου υπάρχει 50-50 εκπροσώπηση και ελπίζουμε ότι τα θέματα του φύλου σε πολυμερές επίπεδο θα είναι όλο ένα και πιο σημαντικά. Θα ήθελα να σας κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση τις ε, διεθνείς εμπορικές σχέσεις αυτή τη στιγμή Μόλις ε, ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση σε τεχνικό επίπεδο μια συμφωνία με τον Καναδά, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει διαπραγμάτευση για τον εξυγχρονισμό της συμφωνίας με το Μεξικό. Πώς πιστεύετε ότι οι πρόοδοι που θα ε, ξεκινήσουν στις διάφορες αυτές συμφωνίες θα επηρεάσουν την ε, συμφωνία με τον Καναδά και πώς μπορεί να αποτελέσει αυτό κίνητρο για να έχουμε συμφωνίες οι οποίες όλο ένα και περισσότερο θα μπορούν να ρυθμίζουν αντιμετωπίζουν τα θέματα της παγκοσμιοποίησης. Πολύ σύντομη ερώτηση από τον κύριο Μποστινάρου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, όπως ε, γνωρίζετε, υπάρχει ένα θέμα πολύ μικρό τεχνικό ίσονο σημασία, αλλά ελπίζω να επιληθεί. Η ρουμανική κυβέρνηση, το ρουμανικό κοινοβούλιο είναι όλοι θετικά διακείμενα υπέρ τη διαδικασία κύρωση. Η αντιπροσωπεία μου δεσμεύεται πλήρω. Μπορούμε να δούμε κάποια πρόοδο. Ο Καναδά θέλει να επενεξετάσει το καθεστώ του ε, των θεωρήσεων διαβατηρίων για του Ρουμάνου και Βούλγαρου υπηκόου, διότι αυτό έχει σημασία εν ώψη και τη διαδικασία κύρωση στο κοινοβούλιο μα. Αυτή ήταν πολύ σύντομη παρέμβαση παρέμβαση πράγματι, κυρία Υπουργέ, για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο χρόνο έχω? 10-15 λεπτά. Λοιπόν, υπήρχαν αρκετές ερωτήσεις. Ο πρόεδρος ε, πρέπει να περιμένει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τον πρόεδρο να περιμένει. Να μην τον αφήσουμε. Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους που ασχολείστε τόσο στενά με αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και πραγματικά πρέπει να πω ότι με εντυπωσίασαν όλες οι επαφές μου με τους ευρωβουλευτές ε, για το πόσο επικεντρωμένοι είστε και πόσο καλά γνωρίζετε αυτή τη συμφωνία. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, ε, διότι ήταν τόσες πολλές αλλά θα προσπαθήσω να σταθώ στα βασικά θέματα και αν υπάρχουν κάποιες απαντήσεις ε, τις οποίες δεν θα δώσω. Ο πρέσβης μας, ο Νταν Κοστέλο, είναι ο πρέσβης του Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πάντα στη διάθεσή σας. Πραγματικά πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για μας, σοβαρά σας το λέω και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα και για τους υπόλοιπους Καναδούς εκπροσώπους να μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Ε, στην αρχή επίση ξέχασα να σα συστήσω κάποιον που γνωρίζετε όλοι, το Στίβ Ριχιούλ, ο οποίο είναι ο επικεφαλή των διαπραγματεύσεων. Ο Μάουρο δεν είναι εδώ, ε. Α, να και ο Μάουρο. Ο διαβόητο Μάουρο. Χαίρομαι πολύ, έχω ακούσει τόσα πολλά για εσά. Είναι ο δικό σα ο διαπραγματευτή. Χαίρομαι που σα βλέπω εδώ και περιμένω να σα μιλήσω αργότερα. Και θα ήθελα επίση πέραν τη ομάδα τη Καναδική κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι και άλλοι Καναδοί εδώ. Ο Μάρκ Μπάρλο από το Συμβούλιο των Καναδών είναι εδώ και νομίζω ότι έχουμε και κάποιους ε, Καναδούς ε, αγρότες ε, και ράντσερς γεωκτήμονες που είναι εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Υπάρχει ένα γενικό θέμα το οποίο έθιξαν αρκετοί εδώ και νομίζω ότι κάποιοι λένε ότι όταν μιλούν οι Καναδοί και οι Ευρωπαίοι θέλουμε να έχουμε ένα τέτα τέτ, αλλά τελικά γίνεται τρίο. Όταν λοιπόν συζητάμε για τον Καναδά, η ευφυΐα e της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης βρίσκεται στο σεβασμό της, ε, και την κατανόηση της ε, κυριαρχίας των κρατών μελών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Καναδάς είναι κυριαρχή χώρα ανεξάρτητη χώρα. Ε, εορτάζουμε την 150η μας επέτειο του χρόνου. Ε, έχουμε μακρά ιστορία ε, ανεξάρτητων αποφάσεων διεθνώς, όχι μόνο σε θέματα εμπορίου. Σας σύστησα το Ταν Κοστάρλο, τον πρέσβη μας, πριν από λίγο και πρέπει να πω ότι συνδέομαι στενά μαζί του γιατί ήταν επιτελάρχης ενός πολύ μεγάλου Καναδά που ήταν και ο μέντοράς μου και προσωπούσε την περιφέρειά μου πριν αναλάβω εγώ, ο Κολ Γκραμ που ήταν και υπουργό Έμεινα ε, όταν λάβαμε την πολύ σημαντική απόφαση να μην συμμετέχουμε στον πόλεμο στο Ιράκ. Είμαστε ανεξάρτητοι, λαμβάνουμε αποφάσει μόνοι μα και αυτό ισχύει και με τι εμπορικέ συμφωνίε. Πρόκειται για συμφωνία μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και οποιασδήποτε άλλη χώρα. Και πραγματικά, εγώ είμαι υπουργό εμπορίου του Καναδά και θα ήθελα να σας ζητήσω να σέβεστε το γεγονός ότι εμείς ερχόμαστε να συζητήσουμε μαζί σας ως ξεχωριστή χώρα. Είμαστε η ενδέκατη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο. Είμαστε χώρα του G7 και να μας ε, μιλάτε αναλόγως. Σας παρακαλώ και ότι και εμείς σας σεβόμαστε αναλόγως. Υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις αναρωτιέστε ε, γιατί μιλάω. Ε, ε, αναφέρθηκα στο θέμα που δεν θέλει να θίξει κανείς. Υπήρχαν ε, πολλές ερωτήσεις για τα θέματα των επενδύσεων. Κάποιες ερωτήσεις μάλλον από πλευρά ε, τη δεξιά, αν χρειάζεται το θέμα αυτό του κεφαλαίου για τις επενδύσεις και μετά ερωτήσατε κατά πόσον είναι αρκετά εύρωστο ώστε να διασκεδάσει τις ανησυχίες ε, των προοδευτικών και μετά μια τρίτη ομάδα ερωτήσεων για το κατά πόσον χρειαζόμαστε καν ένα κεφάλαιο για τις επενδύσεις. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τα απαντήσω όλα αυτά μαζί με ένα επιχείρημα το οποίο είναι αναφανδόν υπέρ του κεφαλαίου επενδύσεων που έχουν ε, αποφασίσει ο Καναδάς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα που με παθιάζει, διότι πρόκειται για πραγματικό επίτευγμα. Είναι ε, παγκόσμια πρεμιέρα διεθνώ και ε, ένας από τους λόγους που υποστηρίζουμε αυτή τη συμφωνία είναι ότι θέλουμε να υλοποιήσουμε αυτό το κεφάλαιο. Γιατί χρειαζόμαστε κεφάλαιο για τις επενδύσεις. Καταρχάς, να επισημάνω το οποίο βέβαια φαντάζομαι ότι θα γνωρίζετε. Εσείς έχετε επινοήσει την ιδέα, ο Μπέρντ και οι συμπατριώτες του ε, σκέφτηκαν ε, το κεφάλαιο για τις επενδύσεις. Το χρειαζόμαστε διότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν είναι πάντα υπό τη δικαιοδοσία ενό εθνικού δικαστηρίου. Υπάρχει μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωση Καναδά και πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει την αρμοδιότητα να κρίνει αγωγέ βάσει της συγκεκριμένη συμφωνίας. Δεν ε, θα είναι πάντα αρμόδιο ένα εθνικό δικαστήριο για να επιλύσει κάθε πτυχή. Αυτό είναι το θέμα. Μπορεί κάποιο να πει ότι υπάρχει ο ΠΟΕ γι' αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να τηρήσουμε τα του ΠΟΕ. Ο Καναδάς έχει μακρά πείρα με τον ΠΟΕΜ. ασχοληθήκαμε με την ίδρυση του ΠΟΕ, πιστεύουμε στον ΠΟΕ, είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι στον ΠΟΕ και χρησιμοποιούμε ε, τακτικά την ε, μέθοδο επίλυσης διαφορών και όπως ξέρετε μία από τις βασικές μας εμπορικές σχέσεις είναι με τους Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι πολύ καλός εμπορικός εταίρος αλλά μπορεί να είναι και πολύ σκληρός εμπορικός εταίρος και θεωρούμε ότι ένα διεθνές όργανο όπως ο ΠΟΕ μπορεί να λύσει διακρίσεις κατά των ε, καναδικών επιχειρήσεων στις Ηνωμένε Πολιτείε, κάτι το οποίο συμβαίνει. Ε, το Δεκέμβριο είχαμε μία απόφαση υπέρ μα ε, στον ΠΟΕ. Το θέμα όμω είναι ότι ο ΠΟΕ είναι ένας μηχανισμός επίλυση διαφορών από κράτος σε κράτος. Ωραία και καλά όλα αυτά, όταν η ε, κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφασίζει μια εσωτερική διαφορά να πάει σε κρατικό επίπεδο. Αλλά από εκεί και πέρα γίνεται πολιτική απόφαση και είναι πολιτικοποιημένη αυτή η διαφορά. Και πρέπει να σας πω ως Υπουργό Εμπορίου ότι κάθε εμπορική επίλυση διαφοράς δεν είναι εποφελία όλων αυτών των διαφορών ε, όταν φτάνουν σε πολιτικό επίπεδο, πολιτικοποιούνται και φτάνουν στις σχέσεις κράτους-κράτους. Αυτή είναι λίγη από τους λόγους που θεωρώ ότι είναι ε, πολύ σημαντικό να έχουμε ένα κεφάλαιο επενδύσεων. Τώρα, για το συγκεκριμένο κεφάλαιο επενδύσεων. Γιατί εγώ ως ε, προεδευτική υπουργό Εμπορίου, γιατί η προεδευτική μας κυβέρνηση το υποστηρίζει με τόσο στένος. Καταρχάς, το δικαίωμα ρυθμίσεων. Το δικαίωμα των ρυθμίσεων είναι ε, εγγεγραμμένο σε αυτό το κεφάλαιο για τις επενδύσεις πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο επενδύσεων. Η συμφωνία μας λέει ρητός ότι ε, απώλεια κέρδους δεν σημαίνει ότι μπορεί κάποιο να προσφύγει στο κεφάλαιο για τι επενδύσει. Επίση, η συμφωνία λέει ρητό ότι τα κράτη έχουν δικαίωμα να αλλάξουν ε, τα, ο καθεστώ επιδοτήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτομάτω μπορεί κάποιο να εκμεταλλευτεί αυτό το κεφάλαιο για τι επενδύσει. Η συμφωνία επίση λέει ρητό ότι η επίλυση ε, διαφορών περί χρέους. Είχαμε κάποια στιγμή το 2008, είναι μια στιγμή περηφάνειας για τον Καναδά και πρέπει να πω ότι οι δικές μας οι τράπεζες δεν χρειάστηκαν ε, εξυγίανση. Επομένως πιστεύουμε ε, στην κυβέρνησή μας. Και είναι όμως κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας ανησυχεί και η συμφωνία λέει ρητός ότι τα θέματα εξυγίανσης χρέους δεν υπόκεινται στο κεφάλαιο για τις επενδύσεις. Άκουσα κάποιες ανησυχίες στο παρελθόν για το κατά πόσον το κεφάλαιο για τι επενδύσεις ε, δεν θα επιτρέψει σε μια χώρα να επιλέξει να θέσει υποκρατικό έλεγχο ένα τομέα ο οποίος μπορεί να έχει ιδιωτικοποιηθεί στο παρελθόν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πρέπει να σας καθησυχάσω εδώ και νομίζω ότι ε, υπάρχουν και κάποιες ε, ανησυχίε από την παλιά συμφωνία επίλυση διαφορών επενδυτή κράτου το δικαίωμα δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων να νομοθετούν διατηρείται στο κέραιό του αυτή τη συμφωνία και μάλιστα είναι γραμμένα με τρόπο το οποίο είναι πολύ σημαντικά και για μελλοντικέ άλλες συμφωνίε. Και κάτι ακόμα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η διαδικασία τη διαιτησία η οποία καθορίζεται βάσει αυτή τη συμφωνία. Και εδώ πραγματικά πρέπει να σα πω ότι ε, φτιάχνουμε κάτι από κοινού, το οποίο είναι καταπληκτικό. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Στη νέα διαδικασία λοιπόν ε, διαιτησίας θα υπάρχουν διαιτητές οι οποίοι θα είναι εκ Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι ε, ασχολούνται με το εμπορικό δίκαιο. Αν θέλει κάποιος να συμμετέχει θα πρέπει να πει ότι εγώ ασχολούμαι αποκλειστικώς και μόνο με αυτό και οι διαιτητές οι οποίοι θα βρίσκονται σε ένα δικαστήριο για να επιλύσουν τα θέματα θα επιλέγονται τυχαία, όχι από, τα, από τους αντιδίκους. Και επίσης θα υπάρχει και μια διαδικασία έφεσης, ένα ε, εφετείο το οποίο οριστικοποιούμε τώρα. Δηλαδή, αντί να έχουμε ένα ε, δικαστήριο, θα υπάρχει κάποιος επικεφαλής ο οποίος θα είναι αρμόδιος για αυτά. Συνειδητοποιώ ότι υπάρχουν κάποιοι εδώ, όπως γίνεται και σε άλλες ε, ομάδες ε, Καναδών, αλλά πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για μια συμφωνία την οποία υποστηρίζουν ε, και το κοινοβούλιο μας και η χώρα. Θα υπάρχουν κάποιοι όμως οι οποίοι δεν είναι υπέρ εμπορικών συμφωνιών, τελεία και παύλα. Και πραγματικά θα ήθελα να σας ε, ε, πω όλους ότι πραγματικά θα ήθελα να υπάρχει ομόφωνη υποστήριξη και στο κοινοβούλιο σας, θα ήθελα να υπάρχει ομόφωνη υποστήριξη και στο δικό μας το κοινοβούλιο, αλλά αυτοί που θέλουν να υποστηρίξουν το εμπόριο και θέλουν να υποστηρίξουν προοδευτικές συμφωνίες, πρέπει να σας πω ότι καλύτερη συμφωνία δεν θα βρείτε και αυτή η συμφωνία θα είναι μια πάρα πολύ καλή ε, συμφωνία που θα αποτελέσει προηγούμενο για προοδευτικές ε, συμφωνίες εμπορίου. Θα αποτελέσει ορόσημο και αν πραγματικά θέλουμε να βελτιώσουμε τα κεφάλαια για τις επενδύσεις, το να τα συζητάμε δεν θα μας οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Χρειάζεται συμφωνία με κάποιον ο οποίος πραγματικά θα εφαρμόσει το σύστημα. Πραγματικά λοιπόν οι προοδευτικοί πρέπει να υποστηρίξουν αυτή τη συμφωνία. Ο Ντέιβιτ ρώτησε για τα θέματα εργασίας και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Εμείς ε, ε, Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για το νέο φορέα ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά σε θέματα εργασίας που συστήνουμε. Εσείς μπορεί να έχετε καλύτερη εμπειρία από αυτού. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη σύσταση αυτού του φορέα. Ε, στη Συμβάση του Διεθνού Γραφείου Εργασία, ο Καναδάς πάντα στην πράξη σε επίπεδο και των 8 συμβάσεων και εδώ θα ήθελα να τονίσω και τον ειδικό ρόλο της κυβέρνησής μου. Εμείς πιστεύουμε στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Δύο από τους πιο πρόσφατους νόμους που πέρασαν και ε, πέντε μήνες είμαστε στην κυβέρνηση ανακαλούν ε, μέτρα κατά των συλλογικών συμβάσεων που είχε εφαρμόσει προηγούμενη κυβέρνηση. Έχουμε επισήμω ε, υπογράψει έξι από τι 8 συμβάσει τη Διεθνού Γραφείου Εργασία. Υπάρχει και αυτή για την παιδική εργασία που ο Στίβ με καθησυχάζει ότι θα έχει υπογραφεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου και θα κυρώσουμε και την 8η. Είμαστε καθοδόν. Άλλε μεγάλε χώρε με τι οποίε έχουμε εμπορικέ σχέσει έχουν υπογράψει μόνο δύο. από τι 8. Για να δείτε τη διαφορά. Τώρα πρέπει να κλείσω, αλλά όχι πριν σχολιάσω το θέμα της Ρουμανίας. Και της Βουλγαρίας βέβαια, εντάξει, μια και είσαστε Ρουμάνους, εσείς όμως είπα τη Ρουμανία. Και συγγνώμη που δεν θα σχολιάσω την Κίνα, θα ήθελα, γιατί ε, εκπροσωπώ την πιο ιταλοπρεπή περιοχή της, του Καναδά, το Τορόντο. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό να πω στους δικούς μου ότι μίλησα και με Ιταλίδα Ευρωβουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα Ιταλικά. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, όπως γνωρίζετε, η, σύμφωνα με τη στρατηγική εταιρική μας σχέση έχουμε δεσμευθεί να απελευθερώσουμε τα ταξίδια ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Καναδά. Είναι, το έχουμε πάρει στα σοβαρά. Ξέρω ότι αυτό δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί στο σύνολό του εξαιτία ε, ε, των θεωρήσεων για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία που υφίστανται αυτή τη στιγμή. Ε, το δουλεύουμε δραστήρια. Ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή γίνονται συναντήσεις. Όπως γνωρίζετε, είμαι υπουργό εμπορίου, δεν είμαι υπουργό μετανάστευσης. Γνωρίζω όμως τις ανησυχίες σας, θα ενημερώσω και τον συναδελφό μου της μετανάστευσης και τον πρωθυπουργό μου και θα τους ε, ε, ζητήσω να εργαστούν για αυτό το θέμα δραστήρια. Και κάτι θετικό τελειώνοντας. Άκουσα από κάποιους. Ε, ένα σχόλιο το οποίο συμμερίζομαι. Αν δηλαδή η Ευρώπη δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον Καναδά και ο Καναδάς δεν μπορεί να συμφωνήσει με την Ευρώπη, με ποιον θα συμφωνήσουμε. Σκεφτείτε το. Σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου ε, είτε η αποτελεσματικότητα των κυβερνήσεων και των κυβερνητικών των κρατικών μηχανισμών. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε, θα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτή η τόσο προοδευτική συμφωνία ανάμεσα στον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που αποτελεί ε, παράδειγμα χάρη στα προοδευτικά μέτρα τα οποία έχει συμπεριλάβει που θα βελτιώσει την ευημερία και στις δύο πλευρές δεν αξίζει να την υποστηρίξουμε εγώ πιστεύω πως ναι Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας που μας μιλήσατε που απαντήσατε στις ερωτήσεις μας στην ταινία, τη Κασαμπλάνκα, η ταινία αυτή τελειώνει με τη φράση «Αυτό αποτελεί την αρχή μιας εξαιρετικής φιλίας». Έτσι θα είναι και για μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ καθίστε. Να περάσουμε στο σημείο 10. Μακροοικονομική χρηματοδοτική βοήθεια προς την την Το έχουμε συζητήσει ήδη μια φορά η ΑΦΕΤ μας ενημέρωσε κατόπιν ότι θα μας στείλει γνωμοδότηση όπως και η Μπούτζ αλλά παρόλα αυτά να δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας την κυρία ε, Ντεσαρνέζ Όπως είπατε το έχουμε δει αυτό το θέμα δεν με ακούτε Je recommence, c'est Όπως υπενθυμίσατε λοιπόν το έχουμε συζητήσει, όλοι γνωρίζουν την κατάσταση στην Τινησία, ας μην τα επαναλάβω. Έχουμε επί μακρόν συζητήσει την εξαιρετικά δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται η Τινησία όχι μόνο εξαιτία τη ε, Συμφωνία Ελεύθερων Ανταλλαγών, αλλά και, το, και εξαιτία των επιγόντων μέτρων για το ελαιόλαδο. Ε, Δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση εξαιτία τη κατάσταση στη Λιβύη, στι πρόσφατε τρομοκρατικέ επιθέσει. Όλοι γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση τη Τινησία έχει λάβει ήδη μακροοικονομική ενίσχυση 300 εκατομμυρίων. Ζήτησαν άλλα 500 εκατομμύρια και γι' αυτό το λόγο συζητούμε τη συγκεκριμένη πρόταση της Κομισιόν. Όπως γνωρίζετε, η Κομισιόν ε, τροποποίησε σε έξι σημεία της την αρχική της πρόταση. Το Συμβούλιο ξαναέδωσε τη σύμφωνη γνώμη του για να μην χάσουμε χρόνο στην παραλογή αυτής της μακροοικονομικής σηματοδοτικής συνδρόμης στην Ισία. Λογικό θα ήταν και εμείς να το λάβουμε υπόψη και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις τροπολογίες για να τελειώσουμε όσο δυνατό πιο σύντομα. Θα ήθελα να πω όμως στην Κομισιόν ότι αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο. Ε, αν η Κομισιόν θέλει να προχωράμε γρήγορα θα πρέπει να προσπαθεί να αποφεύγει να τροποποιεί τα δικά της κείμενα. Γιατί με αυτό τον, αν είχε συμβεί αυτό, η, η ΑΦΕΤ θα είχε τουλάχιστον συντάξει μια γνωμοδότηση και όχι μια απλή επιστολή. Θα είχε πιο πολύ χρόνο. Δεύτερο, δεδομένων των δυσκολιών στις οποίες βρίσκεται η Τινησία, είναι προφανές ότι η συνδρομή αυτή ε, αναμένεται με πολύ αγωνία ε, και θα πρέπει να δοθεί ή πριν λίγο μετά το καλοκαίρι. Ε, μην ξεχνάμε τη Συμφωνία Ελεύθερων Ανταλλαγών, αλλά η εταιρική σχέση με την, την θα πρέπει να λάβει υπόψη τα όσα έχει πει το Κοινοβούλιο για τη Συμφωνία. Δηλαδή θα πρέπει να μην είναι ασύμετρη, θα πρέπει να είναι δημοκρατική διαπραγμάτευση, να, να είναι διαφανής. Και τρίτον, το είπαμε και όταν ήρθε εδώ ο πρέσβης της Τινησίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Τινησία έχει τεράστιο χρέος. Και πολύ καλό να τις ε, δανείζουμε, να την δανείζουμε, αλλά να σκεφτούμε και λίγο πιο καινοτόμες δυνατότητες. Αυτή τη στιγμή το χρέος της φτάνει στο 50% του ΑΕΠ. Την περασμένη φορά που μιλούσαμε με τον πρέσβη, του είπα μήπως σκεφτόμασταν το χρέος ε, να μετατραπεί σε επενδύσεις. Το έκανε η Γαλλία, το έκανε και η Γερμανία. Ε, η... Το Βέλγιο σχεδιάζει το ίδιο. Ίσως στο μέλλον λοιπόν θα ήταν μια δυνατότητα το χρέος να μετατραπεί σε επενδύσεις. Αυτά ως διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντοσαγνέζ. Ισκιώδης. Ο κύριος Σίκο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς ε, συμφωνούμε με τα όσα μας είπε η συγχύτρια. Εξ του ΕΛΚ όμως ε, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτές τις ε, πτυχές γιατί είναι σημαντικό. Το πρώτο, όπου είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, όπως μας ήρθε, τροποποίησε κάποια τμήματα του αρχικού κειμένου το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται σε περίπτωση μακροοικονομικής βοήθειας. Ποιες είναι τώρα οι πτυχές τις οποίες θα ήθελα να σταθώ. <coughs> Καταρχάς, το άρθρο 3, παράγραφος 1 της πρότασης, έχει διαγραφεί η διάταξη βάσει της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει πρωτόκολλο συνεννόησης, το οποίο περιλαμβάνει τις οικονομικές συνθήκες οικονομικής πολιτικής, στην οποία υπόκειται η μακροοικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου και χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες για αυτή την παράγραφο, λογικά, αλλά επειδή ούτε το Συμβούλιο θα καταθέσει τροπολογίε, ε, πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε ούτε το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα όμω να υπενθυμίσω ότι σε γενικέ γραμμέ η διάθεση κονδυλίων ε, για χρηματοοικονομική βοήθεια είναι τμήμα μια σειράς ε, διαρθρωτικών ε, πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που χωρίς αυτά δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Όπως πολύ σωστά είπε η συγγήτρια λοιπόν, δεν θα πρέπει να αλλάζουμε συνεχώς το γενικό κανόνα. Ένα άλλο σημείο το οποίο προέκυψε από τη συνάντηση του ΕΛΚ είναι ότι πρέπει όταν παρέχεται τέτοια μορφής μακροοικονομική βοήθεια ε, η νησία θα πρέπει να ενισχύσει και το ρόλο της ως φίλος και σύμμαχος για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, όπως δεσμεύονται να κάνουν άλλες χώρες της περιοχής. Επομένως, συμφωνούμε με τον κατεπήγοντα χαρακτήρα, συμφωνούμε με τη διάθεση και την τοποθέτηση, αλλά θα θέλαμε να επισημάνουμε κάποιες πτυχές, οι οποίες αφενός ε, αφορούν τις διαδικασίες, δεν μπορούμε να τις ε, ε, ξεπερνάμε συνεχώς και επίσης την ανάγκη να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι πρέπει να υπάρχει και απάντηση ε, και μέσω μεταρρυθμίσεων αλλά κυρίως ε, για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ισιά ο κύριος Λούνς, παρακαλώ. Α, εσείς, παρακαλώ. Ναι, ναι, στηρίζουμε τον εισηγητή. Δεν θα αποβάλουμε τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γκουε. Α, ο Χέλμουτ θα μιλήσει για την Γκουε, αντί για τον κύριο Λεγιάκα. Α, με συγχωρείτε, ξέχασα τη δική μου πολιτική ομάδα. Μα πώς να το πάρω τώρα αυτό, κύριε Πρόεδρε. Να με ξεχνάτε ενώ δεν έχουμε φτάσει ακόμη ούτε στα μέσα της ε, θητείας. Όχι, όχι, δεν θα ερχόμουν στο ΕΛΚ. Ε. Δεν ξέρω πού θα πήγαινα, στο ΕΛΚ δεν θα ερχόμουν. Σοβαρά τώρα. Συμφωνούμε όλοι, τα έχουμε πει πολλές φορές. Πρέπει να κάνουμε πολλές χειρονομίες οικονομικές, διπλωματικές, πολιτικές προς την Τινησία να τη βοηθήσουμε συγκεκριμένα και μακροπρόθεσμα η επίγουσα οικονομική βοήθεια είναι ένα στοιχείο αυτής της προσπάθειας, τα είπε η κυρία Ντεσαγνές. Κάναμε μια συζήτηση για το ελαιόλαδο, υπήρχαν κάποιες ε, διαφορετικές απόψεις. Ξεκινάει μια διαπραγμάτευση, θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς γίνεται. Γιατί ακούσαμε ότι πρέπει να ξαναδούμε τον τρόπο σύναψη συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου, να είναι πιο διαφανής, συμφωνώ, να γίνει και αντινησία, αλλά προβλέπουμε λοιπόν μάκρο χρηματοδοτική βοήθεια 500 εκατομμυρίων που θα πρέπει να εγκρίνει το Κοινοβούλιο για να μπορέσουν να εκταμιευτούν τάχιστα. Η κυρία Ντοσαρνέζ ανέφερε μια ημερομηνία, εγώ λέω τάχιστα. Χαίρομαι που επαναρχόμεθα σε μια αρχή ε, για την οποία ε, θεωρεί η ομάδα μου ότι είναι πολύ σημαντική να ε, εξαρτάται από τη δημοκρατικότητα κάθε καθεστώτος βοήθεια. Αλλά πρέπει να υπάρχει και μια κάποια ευελιξία για αυτήν την αιμονή σε προϋποθέσεις δημοκρατικότητας. Φοβάμαι λιγάκι αυτές τις απαιτήσεις για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να μην πιέζουμε υπερβολικά τους ε, την ίσους φίλους. Ε, τους έχουμε πει ότι ορισμένα πρέπει να γίνουν, αν και ορισμένα έχουν αμφιβολίες επί ορισμένων, να μην επιμένουμε τόσο πολύ. Επανέρχομαι σε αυτά που είπε η κυρία Ντεσαγνές. Η μακροχρηματοπιστωτική βοήθεια είναι μετά. Θα πρέπει να ε, βεβαίως να μας επιστραφεί. Αλλά ήδη είναι μεγάλο το χρέος της Τινησίας. Κάποια στιγμή λοιπόν δεν θα πρέπει να αποφύγουμε, δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε για το τι θα κάνουμε. Θα υπάρξει ε, ελάφρυνση, θα υπάρξει ανακλιμάκωση της αποπληρωμής του χρέους, γιατί αλλιώς όλα αυτά δεν θα είναι παρα παρηγοριά στον άρρωστο. Πρέπει να γίνει συζήτηση. Και με συγχωρείτε που τελικά μίλησα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μορέλ. Ο Χέλμουτ. Θα συνεχίσω προς την ίδια κατεύθυνση. Ο Πατρίκ θα ήθελε να πει και αυτό τα εξή ε, στηρίζει την ανάγκη να βρούμε λύσεις ε, στην πραγματικά περίπλοκη οικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζει την Τινησία. Ιδιαίτερα αυτή τη μεταβατική περίοδο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η χρηματοδοτική αυτή συνδρομή θα ε, είναι απαραίτητη. Το πρόβλημα είναι και πάλι αυτό που συζητούσαμε σήμερα το πρωί με την ευκαιρία της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Ε, το θέμα δεν είναι μόνο για ποιο λόγο ε, δίδονται τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ποια είναι η θέση στην οποία βρίσκεται ο δικαιούχος. Οπότε, αν δίνουμε τέτοια δωρεάν χρηματοδοτική βοήθεια, τότε θα πρέπει αυτή ε, να βοηθάει τη χώρα και να μπορεί η χώρα να την χρησιμοποιήσει. Και θυμάστε τι είχε, πει ο πρέσβης. Είχε πει ότι θα πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα το, ε, το χρέος χρειάζεται περισσότερη βοήθεια με μικρότερα επιτόκια και πιο λαφρείς ε, όρους. Όμως στο μνημόνιο και στην πρόταση της Κομισιόν τίθενται όροι, πρέπει να τίθενται όροι για το τι θα πρέπει να κάνει η χώρα σε ό,τι αφορά τις διαστοτικές μεταρρυθμίσεις. Το είδαμε και με την Ελλάδα. Χρειάζεται να δούμε την πίεση που δέχονται αυτές οι χώρες. Ο κ. Μπροκ, θυμάστε, μας έστειλε μια επιστολή, σας έστειλε μια επιστολή κύριε Λάγκε, και εκεί μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει πίεση χρόνου γιατί έχουμε το Ραμαζάνι και μετά το, Ραμαζάνι έχουμε την καλοκαιρινή, τις καλοκαιρινές διακοπές, οπότε έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ο χρόνος είναι σχετικός μερικές φορές. Ο κ. Ζαντό. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τη σύνδεση ανάμεσα στο Ραμαζάνι και τις διακοπές. Το Ραμαζάνι δεν είναι περίοδος διακοπών. Κάτι τελείως διαφορετικό. Συμφωνώ πλήρως με την κυρία Ντεσαρνές και την έκθεσή της. Ε, είναι επιτακτικό να βρούμε τον τρόπο να βοηθήσουμε την, την Ισία η Ευρώπη έχει μείνει πίσω, έχει καθυστερήσει ε, και σε ό,τι αφορά τι επενδύσει και σε ό,τι αφορά τα ποσά. Ε, βλέπουμε ποια είναι η γεωπολιτική κατάσταση με την γη των την Αλγερία ε, και βλέπουμε ότι αποτελεί δημοκρατικό φάρο ακόμα η Τινησία. Μερικά εκατοντάς εκατομμύρια ευρώ δεν είναι και πάρα πολλά. Οπότε θα πρέπει να είμαστε και πιο γενναιόδοροι. Να σας θυμίσω ότι το 2012 ψηφίσαμε εμείς εδώ ένα ψήφισμα για το χρέος κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Ας το ξαναδεί αυτό το ψήφισμα η Κομισιόν, γιατί εκεί είχαμε ζητήσει από την Κομισιόν να ξαναεξετάσει αυτό το χρέος που είχε συσσωριστεί τις τελευταίες δεκαετίες και μετά έχουμε ένα καινούριο πρόγραμμα βέβαια πιο λαφρύ σε ό,τι αφορά τους όρους του, αλλά και πάλι θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους. Ε, οι όροι του Δούνου του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά και ανθρωπιστικά μέτρα, ε, σίγουρα δεν είναι κατάλληλοι. Δεν θα υποβάλουμε τροπολογία για να περάσει το συντομότερο, αλλά και πάλι νομίζω ότι είμαστε κάτω από τον πύχη. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα Ιταλικά. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να παρέμβω όχι μόνο ως και ε, για την ε, έκθεση που συζητούμε, αλλά και ως εισηγητής για την ε, πολιτική έκθεση ε, την οποία συντάσσω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την Τινησία. Συμφωνώ απόλυτα με τους προλαλήσαντες. Επαναλαμβάνω και εγώ ότι υποστηρίζουμε πλήρως ακράδαντα την ε, δημοκρατική διαδικασία και την ε, ανανέωση της δημοκρατίας στην Τινησία που διαπιστώνουμε τα τελευταία τα, χρόνια. Ε, η βοήθειά μας πρέπει να είναι πλήρης ε, και με ιδιαίτερη ενέργεια. Αναλύοντας τα μέσα τα οποία έχουν διατεθεί, για παράδειγμα στην Ουκρανία, δυστυχώς πρέπει να πω ότι δεν έχουμε κάνει τις ίδιες προσπάθειες. Και αυτό είναι προφανές, λαμβάνοντας υπόψη ότι ναι μεν ε, όσον αφορά το μέσο για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και την ε, μακροοικονομική βοήθεια σε ποσοστό, λαμβάνοντας υπόψη ε, τη δημογραφική κατάσταση της χώρας, έχουμε δώσει κάτι παραπάνω στην Τινησία, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ε, το μέσο για τις ε, επενδύσεις ε, δημοσιοδιωτικό τομέα και όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, να δούμε και τους ε, χορηγούς και τους δωρητές. Επίσης πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα του χρέους που ανέφερε ο συνάδελφος Ζαντό που πήρε το λόγο πριν από σμένα και κυρίως να υπάρχει και η ιδέα ενός ταμείου επενδύσεων κατά την άποψή μου που θα μπορούσε να στηρίξει τους διάφορους τομείς της οικονομίας ώστε να αντιμετωπίσουμε την πολύ μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση. Αν δεν αντιμετωπίσουμε την οικονομική και κοινωνική κρίση κρίση, κατά πάσα πιθανότητα εκθέτουμε αφενός τη χώρα και το λαό στην ε, ρητορική του Ισλαμικού κράτους, ε, ώστε να στρατολογηθούν και αυτοί, και επίσης θα είναι και οπισθοχώρηση. Ε, και θα αντί να υπάρχει δημοκρατία, μπορεί να αποκατασταθεί ένα νέο ε, πολιταρχικό ε, ε, καθεστώς ανα αυτό του Μαγκαλή. Πρέπει λοιπόν να μην επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Επαναλαμβάνω ότι σίγουρα θα υπερψηφίσουμε την μακροοικονομική βοήθεια που συζητούμε τώρα, αλλά θα πρέπει κατά την άποψή μας να είναι και τμήμα ενός πιο συλλογικού σχεδίου. Δεν αρκεί μόνο αυτό, πρέπει να πάμε πολύ παραπέρα και να καταλάβουμε ότι η Ισία πάει πολύ πέρα από τον πληθυσμό της, αν την εξετάσουμε σε βορειοαφρικανικό επίπεδο επίπεδο και σε γενικότερα στον αραβικό κόσμο, διότι μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα ε, για τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Ε, το μόνο θέμα στο οποίο ίσως θα μπορούσαμε να υποβάλουμε κάποια τροπολογία αφορά τον έλεγχο των κονδυλίων που διατίθεται ή πιο συγκεκριμένα την δέσμευση να επιβεβαιωθούν κάποια μέτρα τα οποία αν δεν εφαρμόζονται συνεχώς μπορεί να υπάρχει αναστολή. Υπάρχει αυτό το constantly εδώ το οποίο μας ανησυχεί λίγο γι' αυτό μπορεί να προτείνουμε ε, λίγο πιο αυστηρό ίσως έλεγχο. Ελπίζουμε όμως να μην το χρειαστούμε ποτέ διότι ε, πλέον αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσουμε πλήρη υποστήριξη στην Τινησία περισσότερο από ποτέ και πρέπει να την πιέσουμε να ε, κάνει μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το πλωστάσιο των πόρων που πρέπει να κινητοποιήσουμε για να μπορέσουμε να καταλοπολεμήσουμε την κοινωνική και οικονομική κρίση. Ο κύριος Καστάλτο αυτά. Και τώρα κύριος Ευχαριστώ. Αναφερόμεθα στην βοήθεια προς την Τινησία. Αλλά να θίξω κάτι που δεν έχει ίσως άμεση σχέση αλλά τελικά έχει. Λέμε ότι θα δώσουμε μέχρι 500 εκατομμύρια βοήθεια μέσω δανείων στην Τινησία. Καλό αυτό. Αλλά παράλληλα με τα δάνεια, καλό θα ήταν να δημιουργήσουμε το κατάλληλο κλίμα για να μπορούμε να αγοράσουμε αγαθά και υπηρεσίες. Έτσι θα δημιουργηθεί απασχόληση στην Τινησία αυτό θα βοηθούσε πολύ περισσότερο παρά να τους δώσουμε δάνεια. Τι παράγει η Τινησία και πουλάει στην Ένωση και είναι πολύ σημαντικό για μας. Φωσφορικά μεταξύ του 10 και του 15 ε, μεταξύ 10 και 15 ένα εκατομμύριο μετρικού τόνου ε, εισάγαμε και χρειαζόμαστε αυτό το υλικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι φωσφορική, φωσφορική λύθη, αλλά δυστυχώς πρόσφατα εγκρίναμε ένα νέο κανονισμό για τα νητρικά που σημαίνει μεγάλο περιορισμό για τον, ε, τους φωσφορικούς λίθους αυτούς και κατά συνέπεια θα περιοριστούν πολλοί οι από τη Βόρεια Αφρική συμπεριλαμβανομένης και τη Τινησία. Οπότε, συνοψίζω, βεβαίω να δώσουμε δάνεια στην Τινησία, αλλά από την άλλη μεριά θα σταματήσουμε να αγοράζουμε κάτι που μπορούν να μας πουλήσουν και που το χρειαζόμαστε. Τι έννοια έχουν αυτά. Αυτό θέλω να πω στον εισηγητή. Την εισηγήτρια. Μήπως πρέπει να συντάξουμε μια γνωμοδότηση για το νέο αυτό κανονισμό για τα λοιπάσματα. Γιατί αυτό έχει επιπτώσει στο διεθνές εμπόριο. Μήπως θα πρέπει να το, να το μελετήσουμε. Δεν έχει έννοια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποστινάρου. Όλοι θέλουμε να εκφράσουμε αλληλεγγύη για πολιτικούς λόγους. Γιατί όμως να μην κάνουμε και κάτι πολύ πιο απτό. Η νέα κυβέρνηση της Τινησίας που έχει ευρεία αποδοχή ζήτησε από τις ευρωπαϊκές τράπεζες να την πληροφορήσουν αν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία που έχει κλέψει ο Μπεν Αλή από τον λαό της Τινησίας και να επιστραφούν αυτά στον ε, πραγματικό κάτοχό τους τον λαό της Τινησίας. Δεν αναφέρομαι στο Μοσάκ Φονσέκα, αναφέρομαι σε τράπεζες της Ένωσης. Και καμία ευρωπαϊκή τράπεζα δεν έχει απαντήσει στο αίτημα της ε, κυβέρνησης της Τινησίας. Και δεν τη ζητάνε τίποτα δεν του ζητάνε τίποτα δύσκολο να πούνε ποια είναι αυτά τα προσιακά στοιχεία και να τα επαστρέψουν στην Τινησία στους πραγματικούς κατόχους. Και αυτά που υπάρχουν εκεί είναι πολύ περισσότερα από αυτά που τους δίνουμε. Θα βοηθούσαμε πολύ την οικονομία της Τινησίας και θα αποδείξουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο λόγια. Πρέπει να βρούμε επίσης και ποια άλλα περιουσιακά στοιχεία είναι στην Σαουδική Αραβία που προστατεύει τον Μπεναλή και όταν θα έχουμε την εταιρική σχέση με τη Σαουδική Αραβία τότε εντάξει ωραίο να τους πουλάμε μαχητικά αεροσκάφη να συζητήσουμε και τα λεφτά που έχουν κλέψει από το λαό της Τινησίας. Βέβαια δεν είμαι ονειροπόλος, αλλά πιστεύω ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση μπορούμε να επιτύχουμε πράγματα, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάτι. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς είναι ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος ε, Ταμπάνο. Θα προσπαθήσω να τοποθετηθώ εν συντομία σε σχέση με τα διάφορα σχόλια που έγιναν. Πρώτον, για τον, τη μορφή της βοήθειας, δάνεια, ε, αντί για χρέο και την ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του χρέου. Να πω το εξή: Η κατάσταση του χρέου τη Τινησία δεν είναι δραματική. Ε, οι δείκτε ε, του σχετικοί με το χρέο είναι σχετικά αποδεκτοί σε ό,τι αφορά το επίπεδο και σε ό,τι αφορά τις τάσεις τους. Ε, η τελευταία ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους επιβεβαιώνει την ε, διατρισιμότητα της, των σημερινών τάσεων ε, στην υπόψη του ε, εισοδήματος της ε, χώρας, του κατακεφαλής εισοδήματος. δεν πληρεί ε, τι, τα, τους κανόνες, τους όρους για δωρεάν χρηματοδοτική ενίσχυση η χώρα αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε έχει κάνει και πολύ σημαντική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια τρία-τέσσερα χρόνια για να αυξήσει τη δωρεάν βοήθεια στην Τινησία. Ε, με το πρόγραμμα Ομπρέλα, με το πρόγραμμα για την Αραβική Άνοιξη κλπ. Και ε, όλα αυτά συνδέονται και με τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις προφανώς και έχει κάνει πολύ πρόοδο εκεί, οπότε λογικό να έχει πάρει περισσότερα χρήματα, αλλά έχουμε κάνει προσπάθεια και μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η, του, Τινησία είναι μια από τις βασικές χώρες, δικαιούχιες χώρες ε, για χρηματοδότηση από την ε, ΕΤΕΠ. Σε ό,τι αφορά με την πρώτη της κυρίας Δεσαρνές και άλλων για μια ενδεχόμενη αναρδιάρθρωση ε, του χρέους ή μετατροπή του σε επενδύσεις. είναι κάτι που μπορούμε να το σκεφτούμε, να το μελετήσουμε. το μελετήσουν οι αρχές ε, προσοχή όμως, διότι οποιαδήποτε συζήτηση για αναδιάθρωση χρέους αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, μπορεί να έχει πολύ αρνητική συνέπεια στην πρόσβαση χώρας στις αγορές. Γιατί η χώρα αυτή ακόμα έχει ακόμα ε, πρόσβαση στις αγορές, μπορεί να δανείζεται χρήματα από τις αγορές παρά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Έχουμε ένα εσωτερικό έγγραφο, τεχνικό έγγραφο, το οποίο αναφέρει ότι ε, κατάφερε να δανειστεί ένα δισεκατομμύριο δολάρια στην αρχή του έτους χωρίς σοβαρό πρόβλημα, εντάξει με ψηλό σχετικά επιτόκιο, αλλά διατηρείται η ε, πρόσβαση της αγορές. Τώρα, για την αδειάση του χρέους να πούμε και το εξής. Ε, τα, δάνεια τα οποία δίνουμε είναι δάνεια με πολύ ε, ελαφρύς όρους. Ε, είναι με τους όρους με τους οποίους δανειζόμαστε εμείς από τις διεθνείς αγορές. Πολύ χαμηλά επιτόκια, κάτω του 1% στην πρώτη δόση, για παράδειγμα. Και ε, με ε, αποπληρωμή σε 50 χρόνια. Είναι με πολύ ευνοϊκούς όρους αυτά τα δάνεια, κάτι που βελτιώνει το μείγμα των, του δανεισμού της χώρας. Αυτά είναι τα βασικά που ήθελα να πω για το δάνειο. Τώρα σε ό,τι αφορά το Ραμαζάνι. Αναφέρθηκε και στην ε, ε, επιστολή της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ε, εμείς θα πάμε στην Ισία την επόμενη εβδομάδα για να ξεκινήσουμε συζητήσεις για ένα μνημόνιο. Και ελπίζουμε ότι θα σημειώσουμε πρόοδο τους επόμενους δύο μήνες έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για την υπογραφή της συμφωνίας και την υλοποίησή της ευθύς ε, μόλις οι συνομοθέτες υιοθετήσουν την πρόταση. Σε ό,τι αφορά την ευελιξία, την οποία, οποία ζητήθηκε από την Κομισιόν από ένα συναδελφό σας. Ε, μπορώ να σας πω το εξής. Ήδη ξεκινήσαμε τις, ε, ε εκταμιεύσεις ήδη από τώρα ε, με όρους ε, που αντικατοπτρίζουν αυτό που ήθελαν να κάνουν οι αρχές της νησίας. Έχουμε μια πολύ χαλαρή προσέγγιση στους όρους μας. Από την, από την άλλη μεριά δεν θα βοηθήσουμε την νησία αν καταργήσουμε όλους τους όρους. χρειάζονται όροι γιατί η, την Ισία χαρακτηρίζεται από σημαντικέ αδυναμίε, διαρθωτικές αδυναμίε. Αλλιώ δεν θα την μπορούσαμε να τη βοηθήσουμε αν δεν βάλουμε όρου. Η Αραβική Άνοιξη δεν ήταν μόνο ε, δεν απογοήτευση για το πολιτικό σύστημα, αλλά και για το οικονομικό σύστημα και για το οικονομικό μοντέλο που λειτουργούσε, που εφαρμοζόταν στη χώρα. Οπότε θα πρέπει να τους βοηθήσουμε και στις διαρθωτικές αλλαγές και βέβαια στο να σταθούν στα πόδια τους οικονομικά αυτή τη στιγμή. πρέπει να μην ξεχάσει η χώρα τη μεταρρυθμιστική της ατζέντα. Επίσης, να ευχαριστήσω την κυρία Δεσσαρνές για την έκθεσή της και για την προτάσει τη και για την ε, ε, μη κατάθεση τροπολογιών. Από ό,τι φαίνεται και το Συμβούλιο που κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, έτσι ώστε η πρόταση αυτή να προχωρήσει χωρίς τροπολογίες και να τηρήσουμε τις πιεστικές προθεσμίες που έχουμε μπροστά μας και να βοηθήσουμε την, την Ισία που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Δεσσαρνέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο λόγια. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να είχα ακούσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας λέει ότι αυτό δεν αποτελεί προηγούμενο ε, να ξαναλλάξουμε το κείμενο. Θα με χαροποιούσε και ελπίζω να λάβετε υπόψη αυτό που είπαμε. Ε, καλό θα ήταν να το είχαν πει και αυτοί. Κλείνω η παρένθεση. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη σύγκληση στα όσα ακούσαμε από τους συναδέλφους. Όλοι λένε ότι επήγει η κατάσταση και ευχαριστώ ε, και όλους τους κοιόδης συζητητές που είπαν ότι δεν θα καταθέσουν τροπολογίες ώστε να αποφύγουμε την καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ πολύ όλους λοιπόν. Δεύτερον, όλοι λένε ότι πρόκειται για ένα από τα στοιχεία της αλληλεγγύης που είναι ε, η πιο σημαντική αλληλεγγύη που πρέπει να επιδείξουμε προς την Τινησία γιατί πραγματικά χρειάζεται βοήθεια η Τινησία και στην Τινησία αν βοηθάμε, βοηθάμε τους εαυτούς μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν και δεν θα πρέπει να σταματήσουμε απλώς την μακροοικονομική βοήθεια. Σίγουρα πρέπει να πάμε πολύ παραπέρα και να επιδείξουμε πιο μεγάλη αλληλεγγύη. Ε, τρίτον, όσον αφορά του όρου, ναι, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν δημοκρατικοί όροι, πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Η Τινησία είναι εξαιρετική στην ε, δημοκρατική τη μετάβαση. Δύο λόγια για του όρου για τι ε, διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Η ε, η Κομισιόν προηγουμένως αναφέρθηκε σε χαλαρότητα. Νομίζω ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ εφήγους προσέγγισης και χαλαρότητας. Αυτό το οποίο πρέπει να προτείνουμε στην Τινησία να τη βοηθήσουμε να βρει προοπτική για το μέλλον. Δεν θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις για τις ρυθμίσεις και σας το λέω εγώ, πιστεύω ότι τα θέματα ε, των ε, μεταρρυθμίσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι χρειάζεται να είμαστε νυφάλιοι για να τα διαχειριστούμε αυτά. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βοηθήσουμε και την Τινησία να βρει προοπτική για το μέλλον. Επομένως, απασχόληση, οικονομική ανάπτυξη, οικονομική δραστηριότητα. Εκεί ε, χρειάζεται βοήθεια η την και νομίζω ότι επ' αυτού θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ντεσαρνές. Και τώρα να σας πω την προθεσμία για τις τροπολογίες. 27 Απριλίου, 12 η ώρα. Ψηφοφορία στη συνεδρίαση της 23ης, 24ης Μαΐου. Επειδή είναι εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Εκουαδό, του σημερινού και επειδή Έχουμε άλλα 7 λεπτά μόνο μέχρι την ώρα που ήταν έρθει. Προτείνω να αλλάξουμε τη σειρά των σημείων στην ημερήσια διάταξη, να περάσουμε απευθεία στην ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισημερινού και το κανονισμό να τον δούμε μετά από την ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, καταρχάς Επιτρέψτε μου να σας εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια για τον μεγάλο σεισμό στη χώρα σας. Προτείνω να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή ως ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα του σεισμού. Thanks a lot. Minister, nevertheless, very warm. Παρ' όλα αυτά, να σας καλωσορίσω θερμά, κύριε Υπουργέ, εδώ στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Καλωσορίζουμε και την αντιπροσωπεία σας, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής Ανάπτυξης. Συζητάμε την ε, παράταση της Συμφωνίας ε, Κολομβίας-Περού ε, και Ισημερινού. Έγινε μία αποστολή στον Ισημερινό πριν από μερικές εβδομάδες και πραγματικά προσπαθούμε να προωθήσουμε το ζήτημα και περιμένουμε και την ε, μελλοντική ψηφοφορία για την ε, προσχώρηση του σημερινού στην ε, εμπορική συμφωνία. Εκτιμώ ιδιαίτερα την παρουσία σας εδώ για να συζητήσουμε αυτή τη διαδικασία και από ό,τι γνωρίζω και η Ολλανδική Προεδρία ενδιαφέρεται να επιταχύνει τη διαδικασία. Δεν θα μακρηγορήσω, γιατί είστε ήδη εδώ, να σας δώσω το λόγο. Muy buenas tardes. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο για τα λόγια του και όλη την Επιτροπή για το ένα λεπτό σιγής υπό το φως της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για την ε, άμεση βοήθεια που έστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετά κράτη-μέλη. Ειδικά στην ε, πρώτη φάση έκτακτης ανάγκης και στήριξης ε, του πληθυσμού που έχει πληγεί από το σεισμό του Σαββάτου. Η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη στη χώρα μου. Όμως ε, η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ε, πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προσχώρηση του Εκαδόρ του σημερινού στην υπάρχουσα συμφωνία. Ε, η αντιπροσωπεία μας περιλαμβάνει και ε, ιδιώτες επενδυτές, εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, ε, εκπροσώπους ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανώσεων εργοδοτών και ε, επίσης ε, Ευρωπαίους εισαγωγή προϊόντων από τον Ισημερινό. Όλοι αυτοί ενδιαφέρονται για την υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Ξεκινώντας, θα ήθελα να σας αναφέρω ορισμένα σχετικά στοιχεία για την πρόοδο, σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στη χώρα με τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. Τα τελευταία χρόνια μετά από πλειοψηφία, μετά από απόφαση ε, της πλειοψηφίας, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο προβλέπει ότι η συμμόρφωση με τα ανθρωπινά οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα είναι κακρογωνίως λήθος. Η οικονομία μας ε, είναι από αυτές που πιο γρήγορα αναπτύσσονται, ανα, αναπτύσσονταν, αναπτυσσόταν από το 2007 στο 2015 στη Λατινική Αμερική, περίπου 4% ψηλότερο από ε, το αντίστοιχο ποσοστό άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής. Δυστυχώς ε, ο τελευταίος σεισμός θα επηρεάσει αρνητικά αυτό το ποσοστό, αυτό το δίκτυο. Έχουμε και δύο, άλλες, ε, δύο άλλους όμως εξωτερικούς παράγοντες που μας επηρεάζουν. Και ανταλλάξαμε απόψεις με την Κομισιόν για αυτά τα θέματα και με ορισμένα από τα μέλη του Κοινοβουλίου. Πιο συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια ή τους τελευταίους μήνες είδαμε σημαντική μείωση των τιμών του πετρελαίου. Αυτό είναι πολύ καλό για κάποιες χώρες, αλλά για μας είναι αρνητικό. Γιατί για μας το 2014 ε, αντιπροσώπευε το πετρέλαιο το 52% των εξαγωγών μας. Συνεπώς ε, είδαμε τα έσοδά μας ε, να μειώνονται σημαντικά εξαιτίας της μείωσης του, των τιμών του πετρελαίου. Το άλλο ο άλλο παράγοντα που είναι σημαντική πρόκληση είναι η αύξηση της τιμής του δολαρίου σε σχέση με τα περισσότερα άλλα νομίσματα του κόσμου. Ε, η οικονομία μας είναι οικονομία του δολαρίου. Ε, ε, χρησιμοποιούμε το δολάριο, το οποίο σημαίνει ότι η αύξηση της τιμής του δολαρίου δυσκολεύει τον ανταγωνισμό μας, τον, μειώνει την ανταγωνιστικότητά μας στις διεθνείς αγορές. Μπορώ να σας πω ότι στο σημερινό δεν κάνουμε κοινωνικό dumping. Έχουμε πολύ αυστηρούς εργασιακούς κανόνες, περιβαλλοντικούς κανόνες, τους οποίους ακολουθούμε. Κάτι που σημαίνει βέβαια αυξημένα κόστη στην παραγωγή. Συνεπώς η παραγωγή μας ήδη εξαιτία αυτών είναι λιγότερο ανταγωνιστική από οικονομικής πλευράς και αυτό δυσχεραίνεται εξαιτία της ισοτιμίας του δολαρίου. Είναι δυσκολότερο λοιπόν να ανταγωνιστούμε με χώρες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους αυστηρούς ε, κανόνες ε, με τους οποίους συμμορφωνόμαστε εμείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας από τους ε, στόχους, ένας μεγάλος στόχος του μοντέλου μας ήταν η μείωση της φτώχειας έχουμε μειώσει τη φτώχεια κατά 13 περίπου της 100. Κατά 13 περίπου της 100. Αυτή τη στιγμή το 25% του πληθυσμού μας είναι φτωχό και η εξαιρετική, η, η ακραία φτώχεια έχει πέσει σε μονοψήφια νούμερα, στο 8% το 2015. Αυτό σημαίνει ότι στα 15 εκατομμύρια άτομα που είναι ο πληθυσμό μας, από τα 15 εκατομμύρια, βγάλαμε από τη φτώχεια 1,5 περίπου εκατομμύριο άτομα. Αναμφίβολα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ε, χώρας μας. Αυτή η μείωση της φτώχειας συνοδεύεται και από μια μείωση των ανισοτήτων. Όπως γνωρίζουμε, η μείωση των ανισοτήτων επηρεάζει πάρα πολύ ε, την ανάπτυξη και την καθημερινότητα επίσης, στο βιωτικό επίπεδο. Ε, η ταχύτητα μείωση των ανισοτήτων στο νησιμενό ήταν τρεις φορές μεγαλύτερη από αυτή των υπολείπων χωρών της, Ευρωπαϊ... του, της Λατινικής Αμερικής με συγκεκριμένες πολιτικές. Πολιτικές, κυβερνητικές πολιτικές που αγγίζουν σημαντικές ανάγκες ε, του πολιτισμού μας όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Στην υγεία για παράδειγμα τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε διπλασιάσει, έχουμε διπλασιάσει τον αριθμό των ατόμων ε, τα οποία έχουμε φροντίσει στο ιατροφαρμακευτικό ε, μας σύστημα, το οποίο είναι δωρεάν. Ε, έχουμε κάνει μεγάλες επενδύσεις από το 2007 στο 2015. Τέσσερις φορές υψηλότερη ήταν η ε, ιατρική δαπάνη τα χρόνια αυτά σε σχέση με το παρελθόν. τώρα, στην εκπαίδευση είμαστε αυτοί που πιο πολύ επενδύουμε στην εκπαίδευση στη Λατινική Αμερική σε σχέση με το ΑΕΠ μα. 2% του ΑΕΠ μα πηγαίνει στην εκπαίδευση, στην παιδεία. Υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό όλων των υπολείπων χωρών της περιοχής. Έχουμε μειώσει τον αναλφαβητισμό και σχεδόν έχει μηδενιστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Πέραν όμως των κοινωνικών επενδύσεων, πρέπει να σχολιάσω τι έχει γίνει και με τα εργασιακά δικαιώματα. Υπογράψαμε 61 συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργάνωσης Εργασίας συμπεριλαμβανομένων των 8 θεμελιωδών συμφωνιών. Αυτό δεν έχει καν γίνει από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς το κάναμε. Ο Ισημερινός το έπραξε. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό έχουμε την πιο το πιο χαμηλό δίκτυο ενεργείας στη Λατινική Αμερική. Παρόλο ότι βέβαια οι εξωτερικοί παράγοντες, αυτοί που σας ανέφερα προηγουμένως, το πετρέλαιο και το δολάριο και τώρα ο σεισμός, σίγουρα θα έχουν αρνητική επίδραση στην ε, απασχόληση. Ένα στοιχείο για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι σε ό,τι αφορά τα εργασιακά είναι η καταπολέμηση της παιδικής εργασίας στον Ισημερινό ε, η εργασία των παιδιών ε, ε, από 5 μέχρι 14 ετών έπεσε από το 8% στο 3%. Το 2011 ανακηρυχθήκαμε χώρα που είναι ελεύθερη από παιδική εργασία σε χωματερές. Δεν υπάρχουν πια παιδιά που να δουλεύουν σε χωματερές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρίε. Μόνο 1039 δούλευαν το 2009. Το 2015 έχουμε 90.000 άτομα με αναπηρίες που εργάζονται. Άτομα με ειδικέ ανάγκες ε, που εργάζονται και συνεισφέρουν στην οικονομία μας. Κάτι άλλο που μας κάνει περήφανους είναι η αναγνώριση ε, της ε, μη αμοιβόμενης οικιακής εργασίας. Οι ε, γυναίκες δηλαδή κυρίως που εργάζονται στο σπίτι και τον οποίον ο ρόλος ε, δεν αναγνωριζόταν ε, ούτε θεωρητικά ούτε και οικονομικά, ούτε αμοιβόντουσαν με κάποιο τρόπο, ούτε ανταμοιβόντουσαν με κανέναν τρόπο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ε, αναγνωρίσει αυτό το ρόλο, ε, έχει αυξηθεί ο αριθμός ε, των ατόμων που εργάζονται στο σπίτι δωρεάν και χαίρουν προς κοινωνικής προστασίας. Μετά, ο Ισημερινός είναι μια μικρή χώρα, έτσι, μικρή και για τη Λατινική Αμερική ακόμα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε μια χώρα με μεγάλη πολιτιστική ποικιλία. Με πολυπολιτισμική χώρα θα λέγαμε. Έχουμε ε, επίσης ε, ε, μια πλούσια φύση. Στην, στον Ισημερινό ομιλούνται περίπου 12 γλώσσες και τα περιβαλλοντικά δικαιώματα βρέθηκαν στο κέντρο της δράσης μας. Η το Σύνταγμα μας αναγνωρίζει τα δικαιώματα της φύσης, για παράδειγμα. 1,5 εκατομμύρια εκτάρια δάσους έχουν προστατευθεί με ε, μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση. Καταπολεμούμε δραστήρια την αποψήλωση των δρασών που έχει πέσει κατά πάνω από 50% τα τελευταία 8 χρόνια. Αυτή τη στιγμή η οι προσπάθειες, ε, μάλλον όσα δέντρα χάνουμε από την αποψήλωση, τόσα δέντρα φυτεύουμε περίπου, κατά μέσο όρο Το οποίο σημαίνει ότι ο Ισημερινός βρίσκεται στην πρωτοπορία της προστασίας του περιβάλλοντος. Και να σας πω και ένα ακόμα στοιχείο. Το 2016, το 93% της ενέργειας που θα παράγεται στον Ισημερινό θα προέρχεται από υδροελεκτρικούς σταθμούς. Ε, δεν θα καίμε υδρογονάνθρακες. Θα διατηρήσουμε τα εργοστάσια μας α, για την περίπτωση θα τα χρειαστούμε στο μέλλον, αλλά το 93% της ενέργειας που θα παράγουμε θα προέρχεται από την ίδια τη φύση. Από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως για παράδειγμα υδροελεκτρικούς σταθμούς. Στα έργα αυτά, τα έργα αυτά έγιναν κατόπιν ε, της σύμφωνης του πληθυσμού και κατόπιν διαβούλευση με τον πληθυσμό. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρετε. Γιατί μέσα σε αυτή την κατάσταση εντάσσεται η εμπορική συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό για μας να συνάψουμε αυτή τη συμφωνία, να προσχωρήσουμε σε αυτή τη συμφωνία, ε, η οποία σίγουρα θα φέρει αμοιβαία ωφέλη και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που ήδη βρίσκονται στο νησιμερινό, θα μπορούν ακόμα περισσότερο να έχουν πρόσβαση στη χώρα μας, αλλά ταυτόχρονα θα διατηρήσουμε και εμείς πρόσβαση, θα αποκτήσουμε και εμείς πρόσβαση επίσης όρις με τους γειτονές μας στην ευρωπαϊκή αγορά. Και πιστεύω ότι το διεθνές εμπόριο συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη. Το 30% των εξαγωγών του, του Ισημερινού έχουν ε, ως στόχο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το εμπόριο με την Ευρώπη γεννά δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πολλές σε περιοχές υπαίθρου και πολύ συχνά σε, ε, πρόκειται για ε, θέσεις εργασίας για γυναίκες, ε, όπως για παράδειγμα ε, στην, ε, στον τόνο ή στις γαρίδες. 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν εξαγωγές της, ε, του σημερινού ε, πέρσι που κυρίως από ε, χάρη σε θέσεις εργασίας στις οποίες εργάζονται γυναίκες. Μας ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το κάνουμε ήδη, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί έχει πολύ θετικές συνέπειες σε κάθε τρεις επιχειρήσεις που εξάγουν προς την Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ μικρές ή μικρές ή μέσω επίπεδου επιχειρήσεις. Στις 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα το Εκουαδόρ, όπως ξέρετε, στις 17 Μαρτίου καλύτερα, ε, θίγημεν από το μεγαλύτερο σεισμό στην ιστορία μας, έναν ε, σεισμό 7,8 ρίχτερ. Μέχρι σήμερα έχουμε μετρήσει πάνω από 500 θύματα. Έχουμε θρυνήσει πάνω από 500 θύματα και όσο προχωράμε στη διαδικασία διάσωσης συνεχίζουμε δυστυχώς να βρίσκουμε και άλλα θύματα και άλλους νεκρούς. Έχουμε πάνω από 2.500 τραυματίες και εδώ αυξάνουν συνεχώς τα νούμερα. Σήμερα το πρωί, νωρίς το πρωί, ξημερώματα ώρα Εκουαδόρ, 10 η ώρα, ώρα Ευρώπης, υπήρξε νέος μετασυσμός, 6,1. όπως και ένας προηγούμενος μετασυσμός που ήταν της ε, ιδίας, ε, του ιδίου μεγέθους. Τεράστιες ζημιές έχει υποστεί η οικονομία μας. Ο πρόεδρος Ραφαήλ Κορέα σε μια πρώτη αξιολόγηση έλεγε ότι οι απώλειες από αυτή την καταστροφή σίγουρα θα είναι πολλά δισεκατομμύρια. Και επίσης ε, μην ξεχνάμε ότι το 75% των εξαγωγών του Ισημερινού προέρχονται από τις περιοχές που ε, χαρακτηρίστηκαν έκτακτες ανάγκες μετά το σεισμό. Περιοχές όπου υπάρχει αλληλεία, που υπάρχουν κονσερβοποιίες, κακάο, μπανάνες, γαρίδες, καφέ. Ορισμένοι εδώ ξέρετε τη χώρα μου. Ξέρετε ότι σε αυτή την περιοχή όπου έγινε ο σεισμός παράγεται το 86% των ε, προϊόντων αλληλείας και κονσερβοποίησης εκ των οποίων τα μισά προϊόντα εξάγονται στην Ευρώπη. Παρά την κατάσταση που ζούμε και παρά την ανησυχία που δημιουργεί στην κοινωνία μας, επιλέξαμε να μην χάσουμε το κουράγιο μας και ήρθαμε εδώ για να τονίσουμε ότι μας ενδιαφέρει η διαδικασία διαπραγμάτευσης και ένταξης στην πολυμερή συμφωνία. Δυστυχώς, οι συνθήκες που έχουν προκύψει δεν σημαίνει πως ε, ξεχνάμε ότι ο κόσμος συνεχίζει να λειτουργεί, γι' αυτό δεχτήκαμε την πρόσκλησή σας και ήρθαμε σήμερα. Αλλά θέλουμε να καταστεί σαφές ότι είναι όντως μια εκδήλωση του ενδιαφέροντος της χώρας μου και της δέσμευσης της χώρας μου στη συνέχιση αυτής της διαδικασίας. Και τέλος, η διαδικασία ένταξη στην πολυμερή συμφωνία του Εκουαδόρ έχει πάρει ε, πολύ χρόνο, αλλά θέλουμε να καταλήξει. Είναι σημαντική για την οικονομία μας. Ξέρουμε ότι η καιρή είναι δύσκολη. Έχουμε λάβει τα μηνύματα πολύ καλής ε, θέλησης από διάφορες πλευρές της Ένωσης και είμαστε πεπισμένοι ότι πριν ε, το τέλος του χρόνου θα έχουμε καταλήξει σε αυτήν την εμπορική συμφωνία και θα έχει αρχίσει να ισχύει ότι θα έχει υπογραφεί και ότι θα έχει αρχίσει να ισχύει θα έχει μπει σε εφαρμογή πριν το τέλος του έτους. Και επαναλαμβάνουμε το ενδιαφέρον μας για να προχωρήσουμε σύντομα ε, εντός αυτών των προθεσμιών στην ε, σύναψη αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ Υπουργέ, λέει ο κύριος ε, Πρόεδρος, ε, για, την για την περιγραφή της κατάστασης στη χώρα σας και για την βούληση που εκδηλώσατε να καταλήξουμε τάχιστα στη συμφωνία. Πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στον μόνιμο εισηγητή μας για το θέμα αυτό, τον κύριο Φίσας. okay. Α, πρώτο, ο κύριος Σόλτς. Α, είναι δύο εισηγητές. Πρώτος ο Χέλμουτ, λοιπόν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Υπουργό για την τόσο αναλυτική ενημέρωση. Και είχαμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε για την επίσκεψη του κυρίου Φίσας και μου στη χώρα σας κατά την προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής μας και τονίζω ότι έχουμε πλήρη συνέστηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει το Εκουαδόρ σε αυτήν την τόσο περίπλοκη και λυπηρή κατάσταση. όπως ακριβώς εκφράσαμε μέσω του λεπτού υγιής. Είμαστε στο πλευρό σας. Και πέρα από όλες τις διαπραγματεύσεις, όλες τις συμφωνίες, θα πρέπει να εκφραστεί η ετοιμότητα της Ένωσης να χορηγήσει συμπληρωματική απευθείας βοήθεια αν χρειάζεται. Τώρα επανέρχομαι στην επίσκεψή μας. Το θέμα που μας απασχολεί δηλαδή συμφωνήθηκε στο Κίτο πριν από ένα μήνα ότι ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να εξηγήσετε στα μέλη της Επιτροπής μας του Κοινοβουλίου ποιες είναι οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα σας το οποίο μόλις κάνατε και είναι εντυπωσιακή η περιγραφή της κατάστασης που κάνατε και των εξελίξεων των επιτευγμάτων σας και τονίζω ότι κατά την επίσκεψή μας συναντηθήκαμε με όλους τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησής σας, αλλά όχι μόνο, και με άλλους βουλευτές και χαίρομαι που ο Αντιπρόεδρος της ε, Αρμόδιας Επιτροπής ε, του Κοινοβουλίου του Εκουαδόρη παρευρίσκεται, ακούει την ανταλλαγή απόψεων, συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους ε, του επιχειρηματικού κόσμου και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών αλλά και με μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολείται περισσότερο με την αλληλεγγύη και την κοινωνική πρόοδο στη χώρα σας. Συναντηθήκαμε επίσης με τους αυτόχθονες πληθυσμούς, με εκπροσώπους των αυτοχθόνων πληθυσμών. Συναντηθήκαμε με συνδικαλιστές. Διαμορφώσαμε λοιπόν μια ε, ευρεία άποψη και Όλοι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης τόνισαν την αποφασιστικότητά τους να επεκταθεί αυτή η συμφωνία με τον Περού και την Κολομβία και μέσω της συμμετοχής του σημερινού και υπήρξε πλήρης κατανόηση αυτού που και εσείς είπατε ότι θα είναι θετική αυτή η επέκταση αυτής της συμφωνίας και για τις δύο πλευρές. Είναι λοιπόν προς το κοινό μας συμφέρον. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε συγκεκριμένα τις λεπτομέρειες ούτω ώστε να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες και των δύο πλευρών. Αυτή είναι η ευθύνη του Κοινοβουλίου και γι' αυτό ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε το τελικό κείμενο ούτω ώστε να περάσουμε στη διαδικασία επικύρωσης και την σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου, όπως προβλέπεται με βάση τις αρμοδιότητές μας. Όπως συμφωνήσαμε και την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο Λάγκερ στην συνεδρία της Επιτροπής, συμφωνήσαμε να αποστείλουμε μία επιστολή προς το Συμβούλιο, ούτως ώστε να είναι πλήρως εν γνώση των θεμάτων αυτών που αναφέρατε και το ότι το Κοινοβούλιο είναι πλήρως διατεθειμένο να συμβάλλει ώστε να υπάρξει ομαλή, παραγωγική και επικοδομητική διαδικασία επικύρωση αυτής της συμφωνίας. τη επέκταση τη δηλαδή. Και τονίζω ότι ακούστηκαν και φωνές που εξέφρασαν επικρίσεις που δεν είναι πεπισμένοι ότι το ελεύθερο εμπόριο μακροπρόθεσμα είναι προς το όφελος όλων, αλλά βράχει πρόθεσμα δεν άκουσα κανένα που να λέει ότι δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει στη συγκεκριμένη ε, οικονομική συγκυρία λόγω της κατάστασης όπως την περιγράψατε, λόγω της πτώσης ε, της τιμής του πετρελαίου, καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση για να σταθεροποιηθεί το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον για να υπάρξει βιώσιμη διεύθυνση, ε, να υπάρξει σταθερή ανάπτυξη προς το συμφέρον όλων μας. Ο εισηγητής σε αυτή τη διαδικασία επέκτασης και της διαδικασίας σύμφωνης γνώμης τονίζω ότι έχετε επιτύχει πολλά ήδη που δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί σε πολλές άλλες χώρες της περιοχής και ελπίζω ότι ανταποκρινόμενοι σε όλα τα θέματα που θέτει η διαδικασία επικύρωσης αυτής της επέκταση της συμφωνίας θα μπορέσετε να δώσετε απαντήσεις και σε κάποιες άλλες ερωτήσεις και ε, προσδοκίε από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ και τώρα κύριο Φίσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον αγαπητό Υπουργό και να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή που βιώνει η φιλική σας χώρα, ο Ισημερινός. Ε, εκφράζουμε την πλήρη μας αλληλεγγύη με το λαό του Ισημερινού σε αυτές τις τόσο δύσκολες και σκληρές στιγμές. Ε, ε, δεν ξέρουμε ακριβώς ούτε καν τον αριθμό των θυμάτων αυτού του φρικτού σεισμού. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι συμφωνώ με όλα όσα είπε ο συνάδελφος ε, Χέλμουντ Σόλτς. Να ευχαριστήσω ε, για την εξαιρετική υποδοχή που μας επιφυλάξατε στο ΚΙΤΟ ε, από πλευράς κυβέρνησης. Είδαμε και τον Αντιπρόεδρο, πολλούς υπουργούς, συναδέλφους του Κοινοβουλίου του Ισημερινού. Είχαμε συναντήσεις με την κοινωνία των πολιτών, κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μα. Ίσως πολύ σύντομα θα έπρεπε να επενθυμίσω για κάποιους συναδέλφους πώς έχει κατάσταση ε, για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σημερινού αυτή τη στιγμή. Να επιμείνω ότι στις 31 Δεκεμβρίου του 2014 έληξε η συμφωνία ε, GSP Plus και μετά από το αίτημα του Ισμερινού να συμμετέχει στην πολυμερή συμφωνία με την Κολομβία, το Περού και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπεγράφει μία συμφωνία γέφυρα για δύο χρόνια, ώστε να επιτρέψουμε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις ε, για την ε, ε, συμφωνία. Μπορεί να φαίνεται πολύς χρόνος δύο χρόνια, ε, ο χρόνος όμως περνάει γρήγορα, ξέρουμε ότι υπήρξαν και δυσκολίες και με τις άλλες χώρες των Άνδεων. Ε, δεν ήταν εύκολες οι διαπραγματεύσεις, διότι δεν ήταν μόνο θέμα αποδοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από πλευράς Κολομβίας και Περού έπρεπε να έχουμε αποδοχή. Ε, τελικά καταλήξαμε σε μια τελική συμφωνία και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πλευράς Κολομβίας και Περού και τώρα αυτή η συμφωνία είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, λογικά υπάρχει η συνήθις προθεσμία των τεσσάρων μηνών για να γίνουν οι μεταφράσεις και ταυτόχρονα ε, τα διάφορα νομικά βήματα. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ μεγάλο αυτό το διάστημα αυτή τη στιγμή γιατί ε, δεν επιτρέπεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη συμφωνία πριν από την τελευταία του Ολομέλεια στο Στρασβούργο στις 12 Δεκεμβρίου του 2016. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολλό δε μάλλον μετά την δινή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει το ο σημερινός, ε, να ε, προχωρήσει η συμφωνία. Αυτό είναι θεμελιώδη σημασία, όπως είπε και ο καλός μου φίλος Χέλμουντ Σόλτς και ε, από πλευράς του Προέδρου, του Μπεν Λάγκερ, ε, αποστήλαμε επιστολή στην Ολλανδική Προεδρία ζητώντας από πλευράς ε, της Επιτροπής μας, από πλευράς του Κοινοβουλίου, να ε, περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό αυτή η προθεσμία, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η συνήθις διαδικασία και το Κοινοβούλιο το αργότερο στις 12 Δεκεμβρίου, το αργότερο επαναλαμβάνω, διότι από την επόμενη μέρα θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία. Αν δεν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, ξέρουμε τι προβλήματα θα δημιουργηθούν για το Εκουαδόρ θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η κατάσταση του σημερινού ε, και λόγω των τεραστίων δυσκολιών ε, του σεισμού και τις απώλειες που έχουμε, όχι μόνο σε ανθρώπους αλλά και οικονομικές απώλειες, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές οι εξαγωγές του 30% ε, των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουν χωρίς δασμούς. Διότι πολλοί επιχειρηματίες μας είπαν ότι δεν θα μπορέσουν να αντέξουν να καταβάλουν αυτούς τους δασμούς. Θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ανεργίας, ιδιαίτερα στις ε, παράκτιες πόλεις οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από το σεισμό, όπως πολλοί σωστά μας εξήγησε ο Υπουργός. Εκεί έχουμε και πολύ μεγάλη γυναική απασχόληση, ε, ανήπαντρες μητέρες και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να μην ε, υπάρξει κάποιο πρόβλημα και να εγκριθεί η συμφωνία πριν από το τέλος του έτους. Επίσης, να πω ότι αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει και άλλα πολύ σημαντικά ωφέλη για το Εκουαδόρ. Η οικονομία του Ισημερινού ε, βασίζεται πολύ σε εξαγωγές πρώτων υλών, κυρίως πετρελαίου και με την πτώση του τιμή του πετρελαίου υπήρξαν σοβαρά προβλήματα. Αναφέρθηκε επίσης ε, και τη, η αύξηση της συναλλαγματικής ισοτομίας με το δολάριο και η ε, ενίσχυση του δολαρίου που δημιούργησε προβλήματα και το γεγονός ότι ε, άλλες χώρες εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και αυτό φυσικά δημιουργεί ε, επιπλέον προβλήματα στις σχέσεις με τον Ισμερινό. Η συμφωνία βέβαια θα χρησιμεύσει για να δώσουμε και μια όθηση στη βιοτεχνία και αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό ε, μήνυμα ε, για την ε, προώθηση του Ισημερινού. Σίγουρα το Κοινοβούλιο θα υπερψηφίσει. Δεν θα υπερψηφίσει μόνο τη συμφωνία. Αυτό είναι σαφές και νομίζω ότι θα έχει και μεγάλη πλειοψηφία, αλλά θα επιμείνει για να διευκολύνουμε και στις χρονικές προθεσμίες, ώστε να μπορέσει να υπογραφεί η συμφωνία πριν από το τέλος του έτους δεν εξαρτάται από εμά. Το, πρόβλημα, το θέμα ε, επαφίεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά η διάθεση και ξέρουμε και τι επαφές ε, είχαμε με το Συμβούλιο, ξέρουμε ότι είναι θετική. Ε, επομένως μπορεί να το επιτύχουμε αυτό που είναι και ο στόχος που έχουμε θέσει εμείς αυτή τη στιγμή. Τίποτα άλλο. Να σας ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία σας εδώ ιδίω αυτέ τι τόσο δύσκολε στιγμέ ε, και το γεγονό ότι καταβάλλατε προσπάθεια για να είστε εδώ, δεχόμενοι και την πρόσκληση του συναδέλφου Σόλτ και του υποφαινόμενου όταν επισκεφτήκαμε το Κίτο πριν από κάποιε εβδομάδε. Ευχαριστώ. Κύριε Ζαντή, θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ και πάλι να σα καλωσορίσω κύριε Υπουργέ. Είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων ήδη σήμερα. Για άλλη μια φορά τα θερμά μας συλληπιτήρια για την ε, τραγωδία που έπληξε τη χώρα σας. Και επίσης ε, διαβιβάστε τα συλληπιτήρια και στις οικογένειες των θυμάτων ε, εκ μέρους μας. Ως προς το θέμα που συζητάμε εδώ, να σας διαβεβαιώσω για άλλη μια φορά ότι υποστηρίζουμε αναφανδόν ως πολιτική ομάδα την προσχώρηση του Ισημερινού σε αυτή την εμπορική συμφωνία με την Κολομβία και το Περό. Θα βοηθήσει για να υπάρξει μια όθηση στο εμπόριο, θα βοηθήσει τον ιδιωτικό τομέα και τις επενδύσεις εκατέρωθεν και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από πλευράς Ισημερινού, αυτό θα αποτελέσει πολύ σημαντικό ε, μοχλό για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στη χώρα σας. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα τεχνικά ζητήματα και οι πιθανές καθυστερήσεις για την κύρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να επιληθούν και επίση πιστεύουμε ότι ε, μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα και αυτή η συμφωνία σίγουρα θα τεθεί σε ισχύ στην 1η Ιανουαρίου του 2017. Και φυσικά ακούσατε και από τους άλλους συναδέλφους και βλέπετε ότι υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη και ευρύτερη συνένεση ε, όλο και περισσότερες πολιτικές ομάδες ε, είναι αποφασισμένες να κάνουν ό,τι μπορούν και να ε, μάλιστα όσο πιο γρήγορα γίνεται ώστε να προχωρήσουν τα πράγματα και να άρουμε οποιοδήποτε πιθανό φραγμό ε, για το πρόβλημα αυτό. Σας διαβεβαιώ λοιπόν και πάλι κύριε Υπουργέ ε, ότι εμείς ως ε, ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα εδώ στο Κοινοβούλιο, θα συνεισφέρουμε για να κάνουμε ό,τι μας αναλογεί και να έχουμε ε, την αμοιβαία επιτυχία αυτή, ώστε να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ του Ισημερινού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι με κοινέ προσπάθειες ε, και ε, με τη βοήθεια των άλλων συναδέλφων θα τα καταφέρουμε. Η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ και τα δικά μας συλληπιτήρια και από την ομάδα μου και από μένα την ίδια για τον σεισμό συμφωνώ με τον Χέλμουτ και με τους υπόλοιπους. Ε, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας στηρίξουμε. Σε ό,τι αφορά την εμπορική συμφωνία, η ομάδα μου είναι επικριτική και με την συμφωνία με το Περού και την Κολομβία. Ε, αμφισβητούμε το, τα ίδια πράγματα. Ο, αμφισβητούμε το ότι βοηθά αυτή η συμφωνία στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ε, παλιότερα και το, η σημερινό έλεγε το ίδιο ακριβώ και το ίδιο επιχείρημα ισχυριζόταν το ίδιο πράγμα και η κυβέρνηση άλλαξε γνώμη. Τι ήταν αυτό που την οδήγησε στο να αλλάξει στάση σε ό,τι αφορά το πώς κρίνει αυτή την συμφωνία. Γιατί πιστεύετε ότι αυτή η συμφωνία τελικά θα βοηθήσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Το εμπόριο ασφαλώς και μπορεί να παίξει ρόλο. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς αυτή η εμπορική συμφωνία μπορεί να σας βοηθήσει. Ε, μπορεί για τα βασικά προϊόντα του Περού και της Κολομβίας ε, να αυξήθηκαν ε, οι εμπορικές συναλλαγές, αλλά συνολικά ε, και αν βάλουμε δηλαδή, αν υπολογίσουμε και τα υπόλοιπα προϊόντα, μειώθηκαν για παράδειγμα, αυτό είναι ένα παράδειγμα για το γεγονός ότι η συμφωνία δεν βοήθησε στην οικονομική ανάπτυξη του Περού και της Κολομβίας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε, Υπουργέ, για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ ξεκινώντας με τα συλληπιτήριά μας, πίεση του σεισμού. Μπορείτε να βασίζεστε στη στήριξη του Κοινοβουλίου και της ε, κυβέρνησης της Ισπανίας. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία, νομίζω ότι πλειοψηφικά συμφωνούμε να τεθεί σε εφαρμογή πριν το τέλος του χρόνου. Οι σοσιαλιστές και δημοκράτες ειδικά θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και με αυτό το πνεύμα. Η, το ψήφισμα, στο ψήφισμα μας ε, υπογραμμίσαμε τη σημασία του προγράμματος δράσης και των μέτρων αυτών που ε, συνοδεύουν ε, μια εμπορική συμφωνία. Έτσι ώστε πραγματικά η συμφωνία να στηρίξει την βιώσιμη ανάπτυξη και την βελτίωση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Η χώρα σας έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο, αλλά έφτασε στα αυτιά μου εξής πληροφορία τελευταία σε ό,τι αφορά την, τους περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης. Θα μπορούσατε να μου πείτε ποια είναι η στάση της κυβέρνησης, διότι οι πληροφορίες που φτάνουμε είναι περί περιορισμού, περί περιστολής των ελευθερών. Είναι αληθινές, βάσιμες. Ε, ε, δεν θα... Ε, θα θέλαμε πραγματικά να ξέρουμε αν υπάρχει τέτοιου είδου περιστολή των ελευθεριών. Πρόεδρος. Ο λόγος των Τζοζέπιων ε, από την Εσωτερική Επιτροπή για την ε, κτίμηση των οικονομικών σχέσεων με το Περού και την Κολομβία κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ και εκ μέρου τη Οργάνωση στην Κοινωνία των Πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κόσμο των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, θέλουμε καταρχά να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μα για τα όσα συνέβησαν, ε, κυρίω προ τα θύματα και στι οικογένειε των θυμάτων. Κύριε Πρόεδρε, σε ένα χρόνο από την υπογραφή της συμφωνίας θα πρέπει βάσει κανονισμού να συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης ε, για τα θέματα της συμφωνίας, ε, στην οποία θα συμμετέχουν και μέλη της κοινωνίας των πολιτών και της χώρας σας. Επομένως, ο κόσμος των επιχειρηματιών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ε, και είναι πολύ ευαίσθητο και σημαντικό αυτό που μπορεί να κάνει η κοινωνία των πολιτών, κυρίως και για να διασκεδάσει και τις ανησυχίε που ακούσαμε εδώ στην αίθουσα. Όταν υπάρχουν ασυμμετρίες μεταξύ των δύο ε, πλευρών της συμφωνίας, όταν υπάρχουν πιθανές δυσκολίες, ελοχεύει ο κίνδυνος, οι συμφωνίες, ε, το εμπόριο, οι εισαγωγές και εξαγωγές ε, που μπορεί να προκύψουν. Ε, οι συμφωνίες αυτές από την άλλη πλευρά ε, του Ατλαντικού θα μας βοηθήσουν ε, βέβαια και θα βοηθήσει η κοινωνία των πολιτών να είναι η συμφωνία αυτή επιτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον Ισημερινό. Το ίδιο κάνουμε και με τους συναδέλφους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών του Περού και της Κολομβίας. Ελπίζουμε ότι θα βρεθούν ανεξάρτητες αυτόνομες οργανώσεις που θα μπορέσουν να εγγυηθούν αυτό το έργο. Να σας ευχηθώ καλή δουλειά και να σας πω ότι είμαστε στη διάθεσή σας σε αυτό το στάδιο με την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει μέχρι τούδε από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία με τους συναδέλφους ε, από την Κολομβία και το Περού. Είμαστε πάντα στη διάθεση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ε, των χωρών αυτών και είμαστε και στη διάθεση της κοινωνίας των πολιτών της χώρας σας για να προχωρήσουμε αυτή τη δύσκολη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήρια από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ το λαό του σημερινού και όλοι μα τη συμπαράσταση για αυτά τα τόσο τραγικά γεγονότα. Και εμεί θέλουμε σύντομα να επεκταθεί αυτή η συμφωνία. Το αργότερο τέλος του χρόνου είναι πιο αναγκαίο παρά ποτέ. Πολλές από τις ε, περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό είναι αυτές ε, όπου υπάρχει δραστηριότητα αλίας και θα ωφεληθούν από αυτήν την επέκταση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αρχίσει να ισχύει πριν το τέλος του χρόνου. Άρα και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν ε, τη δουλειά τους έγκαιρα. Το Εκουαδόρ ελπίζουμε Είμαστε πεπισμένοι ότι θα συνεχίσει την εργασία ούτω ώστε να εφαρμοστούν όλα όσα πρέπει να γίνουν για να μπορεί να εφαρμόσει πλήρω τη συμφωνία από 1η Πρώτου 17. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τους υπάρχοντες φραγμούς του εμπόριου και άλλα μέτρα πρέπει να ληφθούν ε, στον οικονομικό τομέα με πλήρη σεβασμό προς όλες τις διατάξεις αυτής της συμφωνίας. Ούτως ή άλλως ε, αυτές είναι υποχρεώσεις της. Είμαστε σε επαφή με την ε, διοίκηση και τον Υπουργό της χώρας. Συνεργαζόμεθα πολύ καλά και έχω την εντύπωση ότι υπάρχει πολύ αξιόλογη πρόοδος. Και εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Η Κομισιόν στις 4 Απριλίου υπέβαλε πρόταση. Κάναμε μια πρώτη συνάντηση στο Συμβούλιο μια πρώτη εξέταση για να συζητηθεί η πρόταση της Επιτροπής. Πήγε καλά. Τώρα θέλουμε να δούμε πόσο σύντομα το Συμβούλιο θα ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ελπίζουμε ότι θα είναι αρκετά σύντομα, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να έχει το χρόνο για να χορηγήσει την σύμφωνη γνώμη, που είναι αναγκαία για να μπορέσει η Επιτροπή να εφαρμόσει ταχαίω τη συμφωνία και ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, θα θέλατε να αντιδράσετε. Καταρχάς, λέει ο κύριο Υπουργό, ευχαριστώ πολύ για την ε, αλληλεγγύη και τα συλληπιτήρια. Η διαδικασία βέβαια αυτή τη στιγμή είναι ενώπιον του Συμβουλίου και είμαστε πεπισμένοι ότι θα το αντιμετωπίσουν με την αναγκαία ταχύτητα λόγω της σημασίας της περίπτωσης και εμείς ως χώρα σε κάθε επίπεδο εργαζόμεθα για να βοηθήσουμε το Συμβούλιο για να συμβεί αυτό. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι οι προθεσμίες ε, ναι μεν είναι περιορισμένες αλλά είναι ρεαλιστικές. Όλα εξαρτώνται από την πολιτική βούληση.

και σε όλες τις δημοσκοπήσεις ε, έχει καταστεί αυτό σαφές. Γιατί ξέρετε ότι στη σημερινή συγκυρία στο Εκουάδωρο, λόγω των εξωτερικών προκλήσεων που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, οι εξαγωγές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Το θέμα πρόσβασης σε διάφορες αγορές είναι πολύ σημαντικό. Και όπως σας είπα, δεν ε, επιδιώκουμε καλύτερες συνθήκες πρόσβασης από τους ανταγωνιστές. Όχι προσπαθούμε να αποκτήσουμε την ισοτιμία. Ισοτιμία πρόσβαση στην αγορά με τους ανταγωνιστές μας. Γιατί είναι σαφές ότι οποιοδήποτε εξετάσει την οικονομία του Ισημερινού θα διαπιστώσει ότι η συμφωνία αυτή είναι πολύ σημαντική για μας. Ορισμένοι, ορισμένα άτομα, ε, ορισμένες οργανώσεις ε, και αυτό είναι απόλυτα κατανοητό, μπορεί να είναι αντίθετη. Οπότε να το συνδυάσω αυτό με το ότι το Εκουαδόρ άλλαξε στάση για ορισμένα θέματα. Αλλά κοιτάξτε, πρέπει να εξετάσουμε τα εξή. Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, οι συνθήκες στις σχέσεις ε, Ένωσης και Εκουαδόρ ήταν σε κάποια φάση υπήρχαν κάποια θέματα ακόμη και εμπορικά. Αυτό ήταν ένα αντικειμενικό λόγο. Αλλά το θέμα είναι ότι έκτοτε έχουν αλλάξει οι συνθήκε. Δεν τίθενται τα ίδια θέματα. Άλλη σημασία έχει μια ε, συμφωνία με την Ευρώπη όταν δεν έχει καμία ανταγωνίστριά μας τέτοια συμφωνία από τη σημερινή συγκυρία που όλε οι ανταγωνίστριε χώρε έχουν μια τέτοια συμφωνία. Πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε στην αλλαγή των συνθήκων στο Εκουαδόρ. Υπάρχει μια αύξηση στις εμπορικές μας συναλλαγές με την Ευρώπη. Είπατε ότι από πλευράς ε, αξίας αλλά και από πλευράς όγκου υπάρχει μια αύξηση. Από πλευράς όγκου ε, πέρυσι είχαμε αύξηση 1,6%. Είναι σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ για τη στήριξη που μας προσφέρατε. Και ακόμη, το θέμα για την ελευθερία έκφρασης δεν μου δημιουργεί δυσχέρειες. Καθόλου. Θέλω να πω στην ε, βουλευτή Ροντρίγκε. Οι εφημερίδε σήμερα, διαβάστε τις σημερινέ εφημερίδες. Ορισμένες ε, επικρίνουν ιδιαίτερα ορισμένα θέματα. Αλλά από αυτό το γεγονό καθίσταται σαφέ ότι υπάρχει δυνατότητα ε, ελεύθερης έκφρασης. Είναι φυσιολογικό βεβαίω να υπάρχει μια διαδικασία, όπως και εδώ, όπως και στις ΗΠΑ, να υπάρχουν νόμοι που να προβλέπουν ε, το σεβασμό της προσωπικότητας των άλλων και ότι η ελευθερία έκφρασης πρέπει να συνδυάζεται με το δικαίωμα στον ιδιωτική ε, σφαίρα και την, το σεβασμό της υπόλοιψης των ατόμων. Μπορείτε να το δείτε αυτό. Διαβάστε τις ε, εφημερίδες μας στο ίντερνετ. Και μπορείτε να δείτε βέβαια και τηλεόραση και ραδιόφωνο να ακούσετε και θα τα διαπιστώσετε όλα αυτά. Για τις ενσυχίες του κυρίου Γιόργενσον για την επικύρωση. Λόγω των εξωτερικών προκλήσεων για τη χώρα μας, χρειάστηκε να λάβουμε ορισμένα οικονομικά μέτρα Ίσως ε, να λάβουμε και άλλα και στο εσωτερικό της χώρας ή και εν σχέση με τις εξωτερικές μας σχέσεις, αλλά τα μέτρα αυτά θα είναι πάντα στα πλαίσια των προδιαγραφών του ΠΟΕ και των κανόνων του ΠΟΕ. Πάντα αυτό κάνουμε και το επαναλαμβάνω. Το, ο Ισημερινός, η κυβέρνησή του, όποια μέτρα και αν λάβει, πάντα θα σέβονται την πολυμερή τάξη και θα σέβονται τους κανόνες του ΠΟΕ. Είναι περίπλοκες οι προκλήσεις ε, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πριν ε, το σεισμό και μετά. Φυσικά ο σεισμός δυσχεραίνει την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Και γι' αυτό η χώρα μου πρέπει να αντιδράσει. Θα χρειαστεί να λάβει μέτρα αλλά πάντα στα πλαίσια του σεβασμού της, της πολυμερούς τάξης, πάντα στα πλαίσια του σεβασμού των κανόνων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Χαρά μας που σας είχαμε εδώ καλεσμένο και συζητήσαμε την προσχώρηση του η σημερινού στην εμπορική αυτή συμφωνία. Κάποιοι συνάδελφοι πάνε να στείλουμε επιστολές στην Ολλανδική Προεδρία για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια